Θα um, ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μας, ε, συνάδελφε. Είμαστε πολύ λίγοι, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Ξεκινώ λοιπόν με την έγκριση της ημερήσιας διάταξη, Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται η μερίστα διάταξη. Τώρα περνάω στο γλωσσικό καθεστώ. Δυστυχώ δεν έχουμε διερμηνία στα δανέζικα, τα μαλτέζικα, κροατικά και τα γκέλικα. Ούτε σήμερα ούτε αύριο λοιπόν διερμηνία σε αυτέ τι γλώσσε. Σε ό,τι αφορά την ε, έγκριση ε, των συστάσεων των συντονιστών με βάση τον κανόνα 205 έχω μία σειρά από διορισμού. Καταρχήν η κυρία Τζιν Λαμπερντ από του ε, Πρασίνου έχει διοριστεί ε, η ε, εισηγήτρια που θα αντικαταστήσει την κυρία Λούνατσεκ που εγκατέλειψε το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την οδηγία για την ισότιμη μεταχείριση. Η κυρία Κάουφμαν ε, από του σοσιαλιστέ έχει διοριστεί εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την πρόταση οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη ε, και την ε, των μέσων πληρωμή άλλων εκτό των μετρητών. Η κυρία Φαζόν έχει διοριστεί εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την ε, προσωρινή ε, ε, επανεισαγωγή των ελέγχων στα σύνορα, στα εσωτερικά σύνορα. Ο κύριο Εμίρια Πάβελ έχει διοριστεί εισηγητή σε ό,τι αφορά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μπαρμπέιντο και την συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Συνότητας και Μπαρμπέντος σε ό,τι αφορά την βραχυπρόθεσμη, τις βραχυπρόθεσμες θεωρήσεις και, το, την απελευθέρωση αυτού του καθεστώτος. Ο κύριος Κον Φερνάντο Λοπέ Αγγιλάρ έχει διοριστεί συγκητρή ε, για την έκθεση ίδια πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τι ανθρωπιστικέ θεωρήσει. Εγκρίνεται λοιπόν αυτέ τι συστάσει ε, ε, των συντονιστών. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε θεωρούμε πω εγκρίνονται. Τώρα από το τρίτο σημείο έχουμε μια ανακοίνωση σε ό,τι αφορά μια σημαντική εβδομάδα, την εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αφρική. Όπω γνωρίζετε, η δική μα Επιτροπή συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην προετοιμασία αυτή τη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αφρική και θα ήθελα οι συνάδελφοι εδώ να ε, παρακολουθήσουν από κοντά όλες αυτές τις ε, δραστηριότητες που θα λάβουν ε, χώρα αυτή την εβδομάδα. Εμείς αύριο θα φιλοξενήσουμε μια ψηλό επίπεδο διάσκεψη ό,τι αφορά την Αφρική στις 22 Νοεμβρίου. Μάλλον θα λάβει χώρα αυτή η διάσκεψη κορυφή εδώ στο Κοινοβούλιο, πέραν από μια ανταλλαγή απόψεω που θα έχουμε εδώ στην Επιτροπή μα αύριο. Οπότε να έχετε κατά νου ότι θα λάβει χώρα και αυτή η διαστήψη κορυφή ε, την Τετάρτη, που είναι σημαντική για τη δική μα Επιτροπή. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τα συστήματα πληροφοριών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στον χώρο τη δικαιοσύνη και των ιστορικών υποθέσεων, θα ήθελα να σα επενθυμίσω ότι μια παρουσίαση σε ό,τι αφορά αυτών των πανευρωπαϊκών συστημάτων πληροφοριών θα λάβει χώρα σήμερα το απόγευμα στι 6.30 μετά δηλαδή από τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Λίμπη, στην ίδια αυτή η αίθουσα, προκειμένου να προετοιμάσουμε την αυριανή συζήτηση που θα κάνουμε σε ό,τι αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα με την Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου υπενθυμίζω, στι 6.30 σήμερα το απόγευμα αυτή η παρουσίαση και στις 6 ώρα σήμερα θα έχουμε και ψηφοφορίες οπότε φροντίστε να έχετε μαζί σας τις ηλεκτρονικές κάρτες για να ψηφίσετε. Τέλος, να εγκρίνουμε και τα πρακτικά ε, της 7 η Σεπτεμβρίου και της 11 η ε, ε, Μαΐου Εάν συμφωνείτε λοιπόν εγκρίνουμε και τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 4 της σημερινής σας διάταξης το οποίο με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω ότι πρόκειται για κοινό σημείο με τα μέλη της ε, Επιτροπής ε, για τη Μεταφορών και της Επιτροπής Αλληλείας. Έχουμε ε, την κυρία Ντάλε, την πρόεδρο δηλαδή, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Να καλωσορίζουμε θερμά και είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε πριν ως μαζί, οπότε πραγματικά την καλωσορίζουμε εδώ θερμά. και ελπίζουμε να προσέλθουν κάποια στιγμή και μέλη από την Επιτροπή Αλληλείας. Πρόκειται λοιπόν εδώ, συνάδελφοι, για μια πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά το project της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής του 2016 και την παρουσίαση έχουμε τρεις εκτελεστικούς διευθυντές εδώ από την αρχή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Συνοριοφυλακή, την ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια τη Θάλασσα και την Υπηρεσία Ελέγχου τη Αλία. Ε, και από εκεί και μετά ε, έχουμε, όπω είπαμε, και μέλη εδώ της, των Επιτροπών μεταφορών και αλληλείας. Ελπίζουμε να προσέλθουν και άλλα μέλη. Σα ζητώ συγγνώμη βέβαια που έχουμε τόσου λίγου παρευρισκόμενου αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι βέβαιο ότι θα αρχίσουν να καταφθάνουν όπως θα καταφθάνουν και διάφορες πτήσεις. Ε, Α ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι και web stream και είμαι βέβαιο ότι υπάρχουν μια σειρά από ενδιαφέροντε οι οποίοι θα παρακολουθούν με ενδιαφέρον και θα ακούσουμε λοιπόν κάποιε παρουσιάσει σε ό,τι αφορά αυτή την πρωτοβουλία. Ε, καλωσορίζω λοιπόν εδώ του ε, κυρίου Λεγκέρη, Σάμπουρε και Μαρκουμίλη και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λεγκέρη Ε, και βέβαια ε, ο κ. Παπέρ είναι ο δικό μα εισηγητή από πλευρά δηλαδή της ε, Επιτροπή. οπότε θα υπάρχει και δυνατότητα να υπάρχουν και κάποια, κάποια σχολιασμοί αυτών των παρουσιάσεων. Α ξεκινήσουμε όμω λοιπόν με την παρουσίαση από την πλευρά του κυρίου Λεγκέρη, του εκπαιδευτικού δηλαδή διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Φυλαξιοσυνών του Ρόντεξ Οπότε, Φαμπρί, νομίζω πώ μπορεί να ξεκινήσει με την παρουσίασή σου, η οποία θα πρέπει να διαρκέσει έω 20 λεπτά. ή μάλλον αφού έχετε συμφανίσει μεταξύ σας, όπως μου είπε μόλις τώρα ο κύριος Λεγκέρη, μπορείτε να αποφασίσετε πώς θα κατανείμετε το χρόνο μεταξύ σας οι τρεις εκτελεστικοί διευθυντές. Άρα ο κύριος Μίλη λοιπόν θα πάρει πρώτο το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν, σας καλωσορίζουμε θερμά στην Επιτροπή μας κύριε Μίλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους Προέδρους των τριών Επιτροπών, ΛΥΜΠΕ, ΠΕΣ και ΤΡΑΜ, που μας κάλεσαν να μιλήσουμε για την συνεργασία των τριών οργανισμών στα πλαίσια του πιλωτικού έργου για την ακτοφυλακή. Είναι σημαντική υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτά που κάνουμε και είμαστε ευγνώμονες στο Κοινοβούλιο που μας επιτρέπει να εργαστούμε σε αυτό το πιλωτικό έργο. Έχουν χρονικούς περιορισμούς, οπότε περνώ στις διαφάνειες και θα ενημερωθείτε από εκεί. Επόμενη διαφάνεια. Πριν από λίγα χρόνια η Κομισιόν έκανε μια μελέτη για τις υπηρεσίες της ακτοφυλακής στην Ευρώπη και στη μελέτη αυτή εντόπισαν 11 δραστηριότητες ως λειτουργίες ακτοφυλακής. έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στη θάλασσα εν μέρη, έχουν να κάνουν με ατυχήματα με τα πλοία, υπάρχει ο έλεγχος των αλλιευμάτων, ε, τελωνιακά θέματα, περιβαλλοντική προστασία, δραστηριότητες τελωνίων και αυτές οι ευρείες δραστηριότητες αντιμετωπίζονται από τις ε, εθνικές αρχές των 28. Έχουμε πάνω από 300 αρχές των κρατών μελών που ασχολούνται με όλα αυτά. Είναι εν μέρη στρατιωτικές υπηρεσίες αλλά και μη στρατιωτικές, πολιτικές υπηρεσίες. Όλες αυτές οι αρχές, πάνω από 300 που είπαμε, στηρίζονται από τρεις οργανισμούς, Frontex, EFCA, EMSA. Συνεργαζόμεθα λοιπόν με όλες τις εθνικές αρχές ε, στα πλαίσια της εντολής κάθε οργανισμού. Έχουμε τον ιδρυτικό κανονισμό και με βάση αυτόν είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμεθα με τις εθνικές αρχές. Και γι' αυτό όντως υπάρχει μεγάλη συνεργασία μαζί τους. Μετά το 2015, πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες ε, μετανάστες ήρθαν από τη Μεσόγειο στην Ευρώπη. Τότε κορυφώθηκε η κρίση του μεταναστευτικού. Και μετά ε, είχαμε το πακέτο για τα σύνορα στο Κοινοβούλιο ε, και το Συμβούλιο. Οι οργανισμοί ρυθμίστηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε να συνεργάζονται ακόμη περισσότερο μεταξύ τους από ό,τι μέχρι τότε. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι εντείναμε τη συνεργασία μας δεν ήταν τίποτε καινούριο αυτό για τους οργανισμούς, γιατί αρχίσαμε να συνεργαζόμεθα ήδη από το 2009 επί τη βάση διμερών και τριμερών συμφωνιών μεταξύ των οργανισμών. Και αυτό το χρονοδιάγραμμα εδώ δείχνει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είχαμε πολλά έργα συνεργασίας μεταξύ των τριών, Frontex, EFCA, EMSA και η τελευταία έγκριση του πακέτου για το, τα σύνορα ε, επισημοποίησε αυτή τη συνεργασία και προσέδωσε και νομική βάση στη συνεργασία αυτή. Αν δείτε εδώ αυτό το πακέτο, αυτή τη δέσμη, βλέπετε ότι περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, ε, επιμερισμένες πληροφορίες, κοινέ πληροφορίε, είναι μεγάλο τομέα. συμμεριζόμεθα ε, πολλές πληροφορίε, γιατί κάθε οργανισμός συλλέγει πληροφορίε διαφόρων ειδών για τη θάλασσα και αυτές είναι κοινέ πληροφορίε μεταξύ των τριών. Ε, ε, υπηρεσίες επιτήρησης, και εδώ υπάρχει μεγάλη συνεργασία. Η ΕΜΖΑ είναι σε σημαντική θέση εδώ γιατί ήδη αρχίσαμε να καταρτίζουμε δυνατότητες επιτήρησης ήδη από το 2004. Ο οργανισμός ε, δημιουργήθηκε το 2 και από τότε αναπτύχθηκαν σειρές διαφόρων δραστηριοτήτων όπου ενισχύσαμε τις ε, ικανότητες επιτήρησης για να συμπεριλάβουμε και νέες τεχνολογίες. Και το ΙΔΕΣΜΙ αυτή μας έδωσε και καινούριους πόρους για να επενδύσουμε στις νέες ε, τεχνολογίες. Δορυφορική παρακολούθηση χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο. Επίσης, μη επανδρομένα σκάφη χρησιμοποιούνται και ε, δίνουμε συμπληρωματικές ε, υπηρεσίες. Η δημιουργία ικανοτήτων είναι σημαντικό κομμάτι αυτής της συνεργασίας, όχι μόνο μεταξύ των τριών οργανισμών, αλλά και με τις εθνικές αρχές. Ε, διοργανώνουν και οι τρεις υπηρεσίες, οι τρεις οργανισμοί, πολλέ, δραστηριότητε πολλές δραστηριότητες εκπαίδευσης ε, των εθνικών αρχών και επίσης επιμερίζονται και οι ικανότητες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης έχουμε και πολλαπλών στόχων ε, επιχειρήσεις όπου γίνεται εντατική συνεργασία των τριών για την επίτευξη καλύτερων ε, αποτελεσμάτων σε αυτούς τους τομείς. Ας δούμε λίγο το πιλωτικό έργο. Προτάθηκε, όπως είπα στην αρχή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2015 και δόθηκαν και πόροι από τον προϋπολογισμό ε, για 18 μήνες. Ο, οι στόχοι του έργου είναι να βελτιώσουν τον συντονισμό και να δημιουργήσουν περισσότερες συνέργειες από ό,τι είχαμε τότε. Βελτίωση της ροής πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών αλλά και μεταξύ των άλλων εμπλεκομένων. Οι, αυτές είναι οι επιχειρησιακές δράσεις στην πράξη. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχε η δυνατότητα να ε, κάνουμε τεστ στην πράξη των δυνατοτήτων μας και έχουμε κοινέ δοκιμές για να βελτιώσουμε και να ενδυναμώσουμε τις δράσεις μας στην πράξη. Οι δράσεις εστιάζουν κυρίως ε, στην κεντρική Μεσόγειο και υπάρχει και συνεργασία στα πλαίσια του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Αυτή είναι η στόχη. Σας διαβεβαιώνω ε, ε, ε, ότι οι στόχοι στα πλαίσια του, του, πιλωτικού έργου έχουν επιτευχθεί. Τώρα, κάποια, κάποιες αρμοδιότητες στα πλαίσια αυτού του πιλωτικού έργου. Πρώτο καθήκον είναι οι κοινέ πληροφορίε, επιμερισμό πληροφοριών. Τι περιβάλλον υπάρχει εδώ. Είναι ένα τεράστιο περιβάλλον. Ε, έχουμε πολλές πηγές συλλογής πληροφοριών από τον τομέα της θάλασσας ε, έχουμε ειδικά για τον χρήστη στοιχεία, για την παρακολούθηση των ε, σκαφών αλλιευτικών και μη μετεωρολογικές πληροφορίες που τις ανεβάζουμε στη βάση δεδομένων μας, ε, συστήματα αυτόματης αναγνώρισης ταυτοποίησης όλων των σκαφών πρέπει να έχουν AIS πομποδέκτη τα σκάφη πάνω από κάποιο τονάζ ε, παρακολουθούμε λοιπόν την κίνηση των σκαφών μέσω δορυφόρου ε, συστήματα απεικόνησης ε, από το 2007 παρακολουθούμε τις περιβαλλοντικές συνθήκες στα ύδατά μας με ε, συστήματα επίσης ε, ε, εντοπισμού και ανείχνευσης δημιουργήθηκαν για λογαριασμό των κρατών μελών από την ΕΜΖΑ συλλέγουμε έτσι στοιχεία για τα ε, σκάφη που φέρουν σημαία της Ένωσης των κρατών μελών. Επίσης έχουμε οπτικές εικόνες δορυφορικές. Αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και δίνει προστιθέμενη αξία στη βάση δεδομένων της ΕΜΖΑ όταν δίνουμε στους πελάτες πληροφορίες. Ε, ε επίσης, ε, πληροφορίες RAPAS ε, ε, έχουμε να, αρχίσει να αναπτύσσουμε αυτές τις πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την κίνηση των σκαφών και παρακολουθούμε έτσι τις υπηρεσίες αυτές. Επίσης έχουμε και το λεγόμενο σύστημα DDS. Αυτές τις πληροφορίες τις μοιραζόμεθα ε, με τους οργανισμούς ΕΜΣΑ και Frontex αλλά και με τις εθνικές αρχές. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών αλλά και με τις εθνικές αρχές. Έτσι ε, προσδίδαμε θέμενη αξία στις αρχές των κρατών μελών και τους Ευρωπαίους πολίτες. Συμπεριλάβαμε αυτό το πορτφόλιο, αυτό το χαρτοφυλάκιο που είναι το ολοκληρωμένο περιβάλλον ε, δεδομένων. Έχουμε συγχωνεύσει όλα τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει σε ένα σύστημα δεδομένων, το οποίο εξυπηρετεί διάφορες αρχές και κράτη-μέλη. Αν δούμε τώρα το αποτέλεσμα αυτού του επιμερισμού πληροφοριών, οι υπηρεσίες ε, των τριών οργανισμών αναβαθμίστηκαν, ε, βελτιώθηκαν, έχουμε πολλές προτεραιότητες ε, σε πιλωτική βάση και τώρα βελτιώνουμε τα δεδομένα τα οποία παρέχονται σε άλλους οργανισμούς. Έχουμε επενδύσει και σε σενάρια υποπραγματικές συνθήκες. Αυτό έχει να κάνει με το τέταρτο το καθήκον και επίσης έχουμε και πολιτική επιμερισμού πληροφοριών και δεδομένων. Είναι μια σαφής πολιτική που υπάρχει εδώ, ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα κλπ. Πάμε τώρα στο δεύτερο καθήκον που είναι η υπηρεσία επιτήρησης. Εδώ επικεφαλής ήταν η Frontex. Θα σας δείξω ένα δίλεπτο βίντεο που έγινε στο Βέλβα εδώ θέλαμε να τεστάρουμε τις υπηρεσίες μας με τις υπηρεσίες Ρέιπας. Δείτε αυτό το βίντεο που είναι δύο λεπτών και δείχνει τι υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε στα κράτη-μέλη και στους διάφορους εμπλεκομένους. to stimulate the cooperation between three agencies to work better in the field of Coast Guard. This is a new initiative which I think is very important and one of our tasks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 Uh, Εδώ βλέπετε την επιτήρηση όσον αφορά τον έλεγχο της, ε, ε, του λαθρεμπορίου. Και τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης. ε, υπόψη τη διαδικασία βλέπετε, διαπιστώνετε ότι η ποιότητα των εικόνων είναι πάρα πολύ καλή. Περιβαλλοντική επιτήρηση. This is search and rescue. Διαδικασίες διάσωσης. Uh, Επίσης ε, κάνουμε και επιτήρηση αλίας. can say that only this drone can fly up to 8 to 10 hours. 8 με 10 ώρες μπορούν να πετάξουν ε, και επομένως ε, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ε, δυνατή διαδικασία επιτήρησης. Αυτό που βλέπετε είναι από ασκήσεις τον προηγούμενο Ιούνιο. Έχουμε πάνω από 100 εκπροσώπους. Έχουμε και έναν εκπρόσωπο και από το Κοινοβούλιο που παρακολουθεί ε, και βεβαίω έχουμε και πολλού εκπροσώπου από τα κράτη-μέλη και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά ήθελα να σα πω. Εγώ ολοκλήρωσα το δικό μου τμήμα και θα δώσω τον λόγο αμέσω στον Φαμπρίς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, αξιότιμους ε, βουλευτές, ε, κυρίως δεν ευχαριστήσω τους τρεις προέδρους των αντιστοίχων κοινοβουλευτικών επιτροπών που μας έδωσαν την δυνατότητα σε μένα και στους συναδέλφους μου να είμαστε εδώ και να σας παρουσιάσουμε το έργο μας. Βρισκόμαστε εδώ ενώπιόν σας διότι ως τρεις οργανισμοί συνεργαζόμαστε και από κοινού παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την σωστή προστιθέμενη αξία που πρέπει να έχουν αυτού του είδους οι διαδικασίες και δραστηριότητες ε, φύλαξης των ε, ακτών. Βλέπετε ταυτόχρονα με την ομιλία μου εδώ αριστερά ένα μικρό βίντεο το οποίο γύρισε ένα ε, μικρό ε, αεροπλάνο το οποίο χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια ενός ε, τυπικού συμβολέου που υπέγραψε η υπηρεσία το 2015 ούτως ώστε να ενισχύσει την δυνατότητα ακτοφυλακής. Ε, ε, αυτό εντάσσεται στο καθήκον 2, υπηρεσία δηλαδή επιτήρηση στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος. Αυτό ε, αυτό το, αυτή η σύμβαση μας έδωσε την δυνατότητα για πάνω από 2.000 ώρες εναέρειας επιτήρησης πάντα στα πλαίσια της ε, δραστηριότητα και της ε, Frontex. Ε, και όσον αφορά συγκεκριμένα το πιλωτικό πρόγραμμα με τις άλλες δύο υπηρεσίες, τους άλλους δύο οργανισμούς, το χρησιμοποιήσαμε για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας μετά από αίτημα της ΕΦΚΑ και ήδη από την Άνοιξη 2017 αρχίσαμε να αναπτύσσουμε αυτές τις δυνάμεις και επίσης είχαμε την ε, δυνατότητα ε, να κάνουμε και πολύ καλές παρατηρήσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της ρήπανσης. Αυτό που είναι καλό να υπογραμμιστεί είναι ότι αυτή η εναέρια επιτήρηση, ε, η FASS, ε, έχει στόχο την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων της εκτοφυλακής και ε, η διαδικασία αυτή έδωσε την δυνατότητα να δημιουργηθεί και ένα νέο είδος κοινή ευρωπαϊκής μονάδας επιτήρησης, monitoring tip, που έχει, που έχει τη βάση της στην Βαρσοβία μέσω αυτού Τών των ομάδων ε, είχαμε εκπώση και άλλων υπηρεσιών, ε, όπω είναι α πούμε ε, θαλάσιων οργανισμών και υπηρεσιών, όσον αφορά την επιτήρηση των ομάδων είχαμε εκπροσώπηση και άλλων υπηρεσιών όπως είναι ας πούμε θαλάσσιων οργανισμών και υπηρεσιών όσον αφορά την επιτήρηση των αλληλευτικών δραστηριοτήτων επίσης σε συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές γιατί δρούμε σε, πολύ κοντά στα όρια της διαδικασίας τρίτων. Επίσης έχουμε εκπροσώπους εθνικών αρχών ε, όσον αφορά και άλλες διαδικασίες ε, ακτοφυλακής και επομένως ε, με αυτές τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες επιτήρησης που βλέπετε και όλες εδώ σε εικόνες καταφέραμε να αναπτύξουμε, την, να, να βελτιώσουμε την δυνατότητα επιχειρησιακής αντίδρασης. Επίσης πριν από κάποιες εβδομάδες καταφέραμε να ε, ε, διαπιστώσουμε 35 περιπτώσεις ανάγκης θαλάσσιας διάσωσης ε, που δεν θα είχαμε την δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε και να ανακαλύψουμε σε άλλη περίπτωση και καταφέραμε να διασώσουμε μετανάστες κυρίως προερχόμενους από την πλευρά της Τινησίας. Στην επόμενη διαφάνεια τώρα Μπορώ να σας πω το εξής. Ε, ε, στα πλαίσια αυτής της ε, συνεργασίας όσον αφορά την, τον επιμερισμό ικανοτήτων, capacity sharing, να σας πω λέω ότι είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις με την υπηρεσία αλληλείας που ζήτησε την βοήθειά μας γιατί η επιχειρησιακή ζώνη ε, της επιχείρησης τρίτων περιλαμβάνει ε, και περιφέρειες ε, οι οποίες αφορούν την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις θαλάσσιες ικανότητες της Frontex αλλά και τις εναέριες ικανότητες έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα η οποία εν προκειμένου θα μπορούσε να βοηθήσει τον έλεγχο των λευτικών δραστηριοτήτων. Συνολικά ε, η Frontex, ε, η ε, Ευρωπαϊκή μαζί με τους άλλους οργανισμούς έχει περίπου 10 σκάφη και ελικόπτερα τα οποία περιπολούν κυρίως στην περιφόρεια της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδος και έχουμε 1.200 συνοριοφύλακες και ακτοφύλακες, 1.200 ε, ε, λέω, στην περιφέρεια της ε, Μεσογείου, που σε κάθε στιγμή έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν και επιπλέον διαδικασίες όπως είναι έλεγχος ελευτικών δραστηριοτήτων ή έλεγχος ρήπανσης περιβαλλοντικής. Ε, και ούτως ή άλλως πληρώνονται ήδη, προβλέπεται το κόστος τους θέλω να πω από, την, ε, από τον προϋπολογισμό. Εδώ βλέπετε ε, ένα σεμινάριο στην Ρώμη στα πλαίσια της κοινής διαδικασίας τρίτων της Frontex αλλά να σας πω επίσης ότι έχουμε και εκπροσώπους εδώ και από την ΕΠΚΑ και από την ΕΜΣΑ. Έχουμε οργανώσει περίπου 20 κοινέ ενημερώσεις, ε, briefing ε, και ε, προέκυψε ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο έτσι ώστε να κατανοήσουν οι εμπλεκόμενοι και το διοικητικό πλαίσιο αλλά και τους στόχους των άλλων οργανισμών γιατί βεβαίως ο κάθε οργανισμός παραμένει στα όρια της εντολής του αλλά υπάρχει μεγάλος βαθμός συμπληρωματικότητας. Εδώ βλέπετε ένα ε, πελίο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της επιχείρησης ε, τρίτων ε, η διαδικασία φόρτωσης εκφόρτωσης αλλιεύματος που πρέπει να επιθεωρηθεί έτσι ώστε να ελεγχθεί η νομιμότητα του αλλιεύματος αυτού και επομένως αυτό εντάσσεται ε, στην ε, συνήθη διαδικασία επιτήρησης. Ε, τώρα, στο επιχειρησιακό πλαίσιο της Frontex προβλέπεται να δίνουμε τέτοιου είδους εικόνες στους συναδέλφους της υπηρεσίας ελέγχου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλίας. Στην επόμενη ε, διαφάνεια βλέπετε κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ ε, βλέπετε μία φωτογραφία την οποία έχει ε, πάρει ελικόπτερο στα πλαίσια του Ποσειδών στην Ελλάδα η Frontex ε, ε, είχε υποψίες ε, για περιβαλλοντική ρήπανση και επομένως άμεσα μετέδωσε τις εικόνες αυτές στους συναδέλφους της ΕΜΣΑ έτσι ώστε να δουν αν και κατά πόσο μπορεί να ανοιχνευτεί η ρήπανση. Επομένως βλέπετε ότι εκμεταλλευόμαστε την ούτως ή άλλως παρουσία του ελικοπτέρου που τόχο και σκοπό είχε την θαλάσσια επιτήρηση ε, σε ελληνικά ύδατα. Εκμεταλλευόμαστε ε, την παρουσία αυτή έτσι ώστε ε, να παράσχουμε μια επιπλέον υπηρεσία προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συγκεκριμένου κράτους μέλους βεβαίως. Στην επόμενη εικόνα βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο η καταπολέμηση, ε, ε, ε, προχωρούμε στην καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας στα πλαίσια συνεργασίας της επιχείρησης Τρίτονα και της επιχείρησης Ποσειδών. Βλέπετε εδώ ένα πλοιάριο το οποίο μεταφέρει ναρκωτικά. Έχουμε συγκεκριμένα μία υπηρεσία συνεργασία, συνεργασίας ε, που ε, μεταδίδει και πληροφορίες ε, στην ΕΜΣΑ. Και βεβαίως υπάρχει και η συνεργασία με τα τελωνία αλλά και με τις αστυνομικές αρχές και τη Europol για να σας δώσω μια εικόνα λίγο πιο συγκεκριμένη όσον αφορά τις κατασχέσεις. Στα πλαίσια της δραστηριότητας της Frontex το 2016 είχαμε 1020 ε, άτομα ε, τα οποία συνελήφθησαν με κατηγορίες ε, διακίνησης μεταναστών, 86 ε, ε, τόνοι ναρκωτικών ουσιών, καθώς επίσης και 14 εκατομμύρια ε, λαθρέα τσιγάρα το 2017. το 2017 είχαμε αύξηση των περιπτώσεων, 156 μέχρι τώρα, οι περιπτώσεις αυτού του τύπου που αντιμετώπισε ε, η Frontex ε, και μάλιστα δύο τρίτα μεταξύ αυτών ε, στην περιοχή μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου. Και για την ώρα έχουν κατασχεθεί 107 τόνοι ναρκωτικών ουσιών. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ένα άλλο παράδειγμα ε, δραστηριοτήτων, κοινών δραστηριοτήτων, ε, υπέρ της διάσωσης. Ξέρετε ότι βάσει του διεθνούς δικαίου ε, υπάρχει υποχρέωση διάσωσης στη θάλασσα και υποστήριξη τέτοιων διαδικασιών διάσωση. Από τον Οκτώβριο του 2016 έχουμε νέα εντολή ε, βάσει των οποίων ε, ε, διαθέτουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τέτοιου είδους διασώσει. Η συνήθι διαδικασία βεβαίω είναι ο έλεγχο των ακτών. Βάσει του ελέγχου όμως αυτού δίνουμε και πληροφορίες στην Ένωση και στην ΕΦΚΑ προτεραιότητα είναι να υποστηρίξουμε ε, ή να διεξάγουμε τέτοιες διαδικασίες διάσωσης ε, που ελέγχονται ε, από το Κέντρο Συντονισμού των Διασώσεων. Στη Ρώμη έχει τη βάση του το, το, Κέντρο Διεθνούς Συντονισμού που προβλέπει βέβαια και άλλες διαδικασίες εκτός από την έρευνα και διάσωση. και αυτό είναι ένα παράδειγμα βεβαίως στην Ιταλία αλλά έχουμε και στην Ελλάδα και στην ε, ε, Ισπανία ε, τέτοιες δραστηριότητες και οι χώρες αυτές συμβάλλουν το 2016 90.000 άνθρωποι διασώθηκαν στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών της Frontex. Το 2017 οι αριθμοί είναι μεγαλύτεροι. 135.000 έχουν διασωθεί ε, στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της Frontex ε, ή ε, και στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος που παρουσιάζουμε σήμερα εδώ. στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε μια άλλη απεικόνηση αυτής, αυτού του επιμερισμού και ανάπτυξης ικανοτήτων ε, βάσει της ε, νέας ε, εντολής αποκτούμε σκάφη μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων leasing στην Ελλάδα το πρώτο σκάφος της, ε, ε, από ε, τους τρεις κοινού οργανισμούς, το βλέπετε και αναφέρει και το όνομα των τριών οργανισμών. Είναι ευρωπαϊκό το πλήρωμα του σκάφους αυτού με 7 εθνικότητες να εκπροσωπούνται στα πλαίσια του, δηλαδή έχουμε ένα είδος πιλωτικού προγράμματος εντός του πιλωτικού προγράμματος ε, και αυτού του είδους η ικανότητα μπορεί εύκολα να ε, μοιραστεί και στο ε, μέλλον έτσι ώστε με την ΕΜΖΑ και την ΕΦΚΑ να έχουμε κοινέ ικανότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι ικανότητες αυτές ως αρχική πλατφόρμα. Βλέπετε λοιπόν ότι η μία υπηρεσία, ο ένας οργανισμός μπορεί να ε, χρησιμοποιηθεί σαν πλατφόρμα για δραστηριότητες ε, άλλων, των άλλων οργανισμών. Εδώ βλέπετε τώρα κάποια από τα διδάγματα εντό εισαγωγικών ε, που έχουμε. Αντλήσει από αυτέ τι εμπειρίε, όπω είπε ο Μάρκο, έχουμε ε, γύρω στις 300 ακόμα και περισσότερες εθνικές υπηρεσίες οι οποίες συμβάλλουν σε αυτές τις ε, εργασίες, σε αυτά τα καθήκοντα της ε, ακτοφυλακής και αυτό που εμείς μάθαμε στο πλαίσιο αυτό του πιλωτικού έργου είναι ότι αυτή η τριμερή συνεργασία, αυτές οι κοινέ δράσεις, δηλαδή ΕΦΚΑ, ΕΜΖΑ και Frontex έχουν βοηθήσει και τα ίδια τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τι επιτυχάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι δεν επιτυχάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι εδώ δεν είχαμε να κάνουμε εικονικό περιβάλλον, είχαμε να κάνουμε πραγματικέ δράσει, οι οποίε έλαβαν χώρα σε πραγματικό χρόνο. Και ε, κάτι τέτοιο βέβαια είναι και αποδοτικό, αποτελεσματικό από πλευρά κόστου, γιατί όπω βλέπετε και με βάση τα αποτελέσματα εδώ, ήμασταν σε θέση να αναλάβουμε δράση σε μια σειρά από διαφορετικού τομεί τη νομοθεσία, αλλά πάντοτε βέβαια η κάθε υπηρεσία στο πλαίσιο τη εντολή τη. Σα ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον συνάδελφο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Προέδρους των τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών ε, Αλίας, Λίμπε ε, και ε, Τραν για αυτήν την συνάντηση. Όπως είπαν και οι τη συναδελφοί μου, ένα σημαντικό στοιχείο ε, του ε, πιλωτικού προγράμματος αφορά τη συνέργεια και την ε, δυνατότητα αλληλεπίδρασης και διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών. Εδώ βλέπετε ας πούμε δεξιά ταυτόχρονα επιτήρηση των ακτών και διάσωση στην ίδια περιοχή. Ε, στο δεξί τμήμα της διαφάνειας βλέπετε το sighting αυτού του είδους ε, ε, της δραστηριότητες ανείχνευσης βάσει της Frontex. Αυτές είχαν εξαιρετικά σημαντικό αποτέλεσμα και όσον αφορά την επίπτωση και την επίδραση που μπορεί να είχαν για τις αλλιευτικές δραστηριότητες. Ε, απ' την άλλη πλευρά ε, ε, βλέπουμε και η υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας που ε, ταυτοχρόνως εξυπηρετείται. Ε, θα ήθελα να πω ότι η διαλειτουργικότητα ε, επίσης της εναέριας επιτήρησης ήταν πάρα πολύ σημαντική και όσον αφορά τα αποτέλεσματα που μπορεί να έχει και που είχε για τον έλεγχο της αλίας. Μας ενδιαφέρει βεβαίως ιδιαίτερω η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, γιατί δεν μας ε, ε, ενδιαφέρει μόνο να συνεργαζόμαστε και να συντονιζόμαστε μεταξύ μας, μας ενδιαφέρει να παρέχουμε μια σωστή υπηρεσία στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να σας πω ότι είχαμε την ε, δυνατότητα να κάνουμε πολύ ε, ενδιαφέρουσες μικτές αποστολές ελέγχου συνόρων αλλά και ταυτόχρονα ελέγχου αλληλευτικής διαδικασίας. Όσον αφορά τώρα έναν απολογισμό για το καθήκον 4, μπορώ να πω τα εξής. Είχαμε πέντε ε, επιχειρήσεις ε, ε, ελέγχου της αλίας μέσω πλοίων της σκαφών της Frontex. Βεβαίως εμείς συμμετείχαμε και σε κοινέ δραστηριότητες στα, πλαίσια του Ινταλό στην Μεσόγειο και στην Δυτική Μεσόγειο και Ποσειδών στην Ανατολική Μεσόγειο οι δραστηριότητες ε, ε, τύπου ε, sightings ήταν 76 στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον. Τον Μάιο του 2017 ε, είχαμε επίσης ε, μια ε, ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία και ανάπτυξη ε, σχεδίου που έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την ε, αλληλεία, κυρίως μέσω δορυφορικής επιτήρησης. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ε, στην, στο τρίτο καθήκον που είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων εμείς ε, συμμετείχαμε ε, σε διαδικασίες ε, κατάρτισης καθώς και διαδικασίες δημιουργίας περιεχομένου. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένας κοινό πίνακας αναφοράς επί θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και που μπορεί να έχουν επίπτωση στις ελληνικές δραστηριότητες. Προχωρήσαμε σε χαρτογράφηση λοιπόν οργανισμών και των υπηρεσιών που μπορεί να έχουν κοινού στόχους. Ε, είδαμε και αναλύσαμε τις υφιστάμενες ε, συμφωνίες οι οποίες μπορεί να έχουν ε, καλή επίπτωση σε αυτήν την οικοδόμηση ικανοτήτων. Είχαμε λοιπόν κατάρτιση ε, και των δικών μας ε, μελών αλλά και εκπροσώπων ε, του προσωπικού που ασχολείται με τα θέματα αυτά στις χώρες μέλη έτσι ώστε να δημιουργηθούν καλές διαδικασίες εκπαίδευσης και ένα, μια ικανή ποσότητα πληροφοριών έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει μια σωστή διαλειτουργικότητα μεταξύ του προσωπικού των διαφόρων υπηρεσιών Όσον αφορά την, αυτή την δράση 3 της ε, ΕΦΚΑ, μπορώ να πω ότι ε, σε συνολικό ε, επίπεδο είχαμε μια καλή παρουσία όσον αφορά και συμβολή, όσον αφορά την δημιουργία κοινών ικανοτήτων, επιτήρησης, κατάρτισης προσωπικού, ανταλλαγής προσωπικού και διαλειτουργικότητας του προσωπικού. Οδηγούμε λοιπόν τώρα ε, να εξάγω κάποια συμπεράσματα, μάλλον εγκάρσια όσον αφορά αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Θα έχετε διαπιστώσει ίσως ότι λίγες ε, δραστηριότητες ε, του πιλωτικού προγράμματος αφορούν τις μικτές δραστηριότητες. Επίση, ε, αναφερόμαστε και σε διαδικασίε ε, οι οποίε ε, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκπροσωπείται μέσω τη Κομισιόν αλλά αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι σημαντικό στα πλαίσια αυτά να δημιουργήσουμε διαδικασίε οι οποίε θα αποφύγουν τι επικαλύψει και οι οποίε θα ενδυναμώσουν τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τι ομάδε μα, οι οποίε έδειξαν ιδιαίτερη μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής ε, και για μία ακόμα φορά ε, ενδυναμώνεται και η ε, ιδέα ότι μέσω της συνεργασίας μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να χρησιμοποιηθούν ταυτοχρόνως καλύτερα οι ευρωπαϊκοί πόροι. Όσον αφορά τώρα την επιμήκυνση του πολιτικού προγραμμάτου προγράμματος ε, ε, η συνεργασία αυτή ε, θα ενδυναμωθεί. Εκτός από τους τέσσερις αρχικούς στόχους που αφορούν την διαχείριση, την ικανότητα, την αύξηση ικανοτήτων προστίθεται και η διαδικασία ανάλυσης κινδύνου που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντική. Διοικητική συνεργασία επίσης έχει ξεκινήσει έτσι ώστε με συμβατικό τρόπο ε, να προχωρήσουμε ε, σε μια συνεργασία η οποία θα διαθέτει ε, μια σύμβαση πλαίσιο επίσης μια ρύθμιση τριμερούς, μια μάλλον τριμερής ρύθμιση εργασίας προϋποθέτει και προβλέπει παρόμοιες ε, διαδικασίες ε, ε, για, τα διοικητικά συμβούλια των τριών οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε καλύτερα να παρακολουθούμε σε ετήσια βάση τον ρυθμό της συνεργασίας των τριών οργανισμών. Βάσει των αρμοδιοτήτων που τους έχουν δώσει οι συνομοθέτες ε, έχουν την δυνατότητα οι τρεις υπηρεσίες να συμβάλλουν ε, στην επιτήρηση των συνόρων, των ακτών ε, αλλά και των αλευτικών διαδικασιών και βεβαίω ε, προβλέπεται και η οργάνωση, η διοργάνωση ε, ε, πολλών εκδηλώσεων όπω είναι το φόρουμ του Απριλίου του 2018 που θα ενισχύσει την συνεργασία. Δεν πρέπει να λησμονούμε βεβαίω εν μέσω όλων αυτών των διαδικασιών ότι εδώ και μέσω αυτών των αποστολών εξυπηρετούμε και υπηρετούμε του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους τρεις εκτελεστικούς διευθυντές ε, ε, αυτές τις παρουσιάσεις ε, που ήταν πολύ ζωντανές. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά θέλω να διασφαλίσω ότι τα μέλη της Επιτροπής μας τα οποία σας άκουσα με προσοχή και συμμετέχουν σε αυτές τις εργασίες έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα που θέλουν. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον κύριο Πάμπριξ ο οποίος ήταν ο εισηγητής μας ε, σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα τη ε, συνολοφυλακής και βέβαια θα δώσω το λόγο στη συνέχεια στην κυρία Αντέλη από την πλευρά τη ε, Επιτροπής Τραν και από εκεί και μετά υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι όπω ο κύριο Στίβενς Γκρίσμπεκ και άλλοι. Κύριο Πάξης λοιπόν καταρχήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους αξιότιμους διευθυντές που βρέθηκαν σήμερα εδώ και μοιράστηκαν μαζί μας αυτές τις πληροφορίε, παρότι βέβαια ε, κάποιοι ακόμα συνάδελφοι δεν έχουν προσέλθει γιατί ακόμα γιορτάζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και εγώ θα ήθελα λοιπόν να σα ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που είχα να συμμετάσχω ε, στο workshop που διοργανώσατε στι αρχέ του καλοκαιριού στη Λισαβόνα γιατί εκεί είχαμε ε, τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Διακόπτει ο πρόεδρος τον κύριο Πάμπρεξ υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο, κάποια παράσιτα. Ξανά ο κύριο Παύρεξ. Ναι, πρόεδρε, θα συνεχίσω πολύ γρήγορα, ε, γιατί ξέρω ότι βρισκόμαστε το πίεση χρόνο. Άρα λοιπόν διαπιστώνω ε, σε ποιο βαθμό είναι απαραίτητο να υπάρχει μια αλληλεπικάλυψη και συμπληρωματικότητα των εργασιών μεταξύ αυτών των τριών ε, υπηρεσιών ε, Frontex. Τρία ερωτήματα θα ήθελα να θέσω από τη δική μου πλευρά. Το πρώτο ε, αφορά στο ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποιο είναι το συμπέρασμα. Δηλαδή, ο τελευταίο εκτελεστική διευθυντής αναφέρθηκε ε, λίγο πολύ σε αυτό, αλλά ποιο είναι το επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Γιατί, βέβαια, σε τελική ανάλυση αυτά τα ζητήματα παραμένουν εθνική αρμοδιότητα. Οπότε, αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών, αυτή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτιών μπορεί πράγματι να μεταφραστεί σε απτά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την, ε, ε, το, την εμπορία ανθρώπων, σε ό,τι αφορά την ε, διακίνηση λαθρομεταναστών, σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο και οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, α, αυτά τα ερωτημάτα μας οδηγούν στο γενικότερο ερώτημα του, του, νομικού πλαισίου, πράγμα βέβαια το αποτελεί ε, και δική μας αρμοδιότητα, της Επιτροπής μας και γενικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε λοιπόν κάποια πρόταση ε, προς εμάς ως προς το πώς να βελτιώσουμε την ομοθεσία προκειμένου τα διδάγματα που αντλήσατε από αυτούς τους 18 μήνες από αυτό το πιλωτικό έργο θα μπορούσαν να να, επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχει κάποιος τρόπος για να ε, μέσω της νομοθεσίας να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί βέβαια ε, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με συνεργασία. Με αυτά τα έργα δημιουργούμε και περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ μας, ε, τη καλύτερη συνεργασία. Ναι, έχετε δίκιο, δηλαδή ε, τα σχέση είναι σημαντική μεταξύ αυτών των υπηρεσιών και βέβαια ειδικότερα ε, η υπηρεσία τη ΕΜΣΑ ε, μπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητα τη Επιτροπή Μεταφορών. Οπότε δίνω το λόγο στην πρόεδρο τη Επιτροπή Μεταφορών, την κυρία Ντέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Κλοντ. Είναι μεγάλη χαρά που έχουμε εδώ μαζί μας τους εκτελεστικούς διευθυντές των τριών ευρωπαϊκών οργανισμών που έχουν αποδείξει ότι μπορούν όχι μονάχα να συντονιστούν και ότι δεν χρειάζεται απλό συντονισμός, αλλά χρειάζεται στενή συνεργασία έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για την Ευρώπη. Όταν σκεφτόμαστε ε, και όταν αναλογιστούμε ότι είναι πολλοί οι μετανάστες οι οποίοι μέσα από πολύ επικίνδυνους δρόμους και με κίνδυνο της ζωής τους εξεκολουθούν να περνούν την Μεσόγειο, οφείλουμε να σκύψουμε σοβαρά πάνω από το πρόβλημα αυτό ε, γιατί η παρούσα κατάσταση επηρεάζει και την εργασία αλλά και τον ρόλο που έχουν ε, οι ε, διάφοροι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερος δε αυτούς με τους οποίους συναντώμεθα σήμερα. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών Πρέπει να πω ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ε, τον, ε, την εργασία τη, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και χαίρομαι ε, που ο, εκτελεστικός της διευθυντής, τον οποίο συχνά έχουμε ακούσει στην δική μας επιτροπή, είναι σήμερα εδώ. Πραγματικά ο ρόλος της είναι σημαντικός. Ε, έχει καταφέρει να ελέγξει όντως την ε, ασφάλεια στη θάλασσα, αλλά και να παράσχει και κάποιες αρχές βάσει ε, των οποίων μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική η ασφάλεια στην θάλασσα. Πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος διαρκώς ε, εξελίσσεται. Αναθεωρήθηκε πέντε φορές ε, μάλιστα ε, η εντολή του οργανισμού αυτού με νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα στο πλαίσιο κάθε ανανεωμένης εντολής και βεβαίως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την ΕΦΚΑ. Πιστεύω ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε, να ενισχύσουμε την ε, ε, ικανότητα ε, τις ικανότητες μάλλον που έχουν ε, οι οργανισμοί αυτοί και την ικανότητα της, Ευρωπαϊκής, ε, της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής γιατί δεν είναι ικανά τα κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τι μπορεί να γίνει όσον αφορά το θέμα αυτό στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, μέχρι τώρα το πιλωτικό πρόγραμμα μας έχει δώσει καλά αποτελέσματα, αντίστοιχα με τους στόχους που είχαν τεθεί. Ε, το είπατε, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε η χρήση νέων τεχνολογιών και νέων συστημάτων όπως είναι ε, τα μη επανδρομένα ε, αεροσκάφη, τα drones ε, ή όπως είναι τα προγράμματα Κοπέρνικους δίνουν την δυνατότητα για πιο ολοκληρωμένη επιτήρηση και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή συζητούμε την ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, ε, ε, για τις αεροπορικές μεταφορές ε, και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να μας απασχολήσουν αντίστοιχοι προβληματισμοί όπως ας πούμε ε, το θέμα της ε, χρήσης ή της απελευθέρωσης πετρελαίου καυσίμων σε περίπτωση ας πούμε που υπάρχει κάποιο πλοίο σε κίνδυνο. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε και να διασώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αγαπητέ Κλοντ, είναι πάρα πολύ σημαντικό που εδώ ε, ε, συνεδριάζουν όχι μόνο, μόνο από κοινού τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, αλλά και οι εκτελεστικοί διευθυντές τριών ευρωπαϊκών υπηρεσιών ιδιαίτερα σημαντικών. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και αποτελεί ένα καλό παράδειγμα συνέργειας. Θα πρέπει να υπάρχουν συνέργειες όμως και με τις εθνικές αρχές γιατί δεν πρέπει να τις λησμονούμε. Μερικές φορές μας δημιουργούν προβλήματα, προσκόμματα αυτές οι εθνικές αρχές. Δεν πρέπει να το κρύβουμε. Ε, εύχομαι λοιπόν να έχει καλή πορεία ε, η Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εκτοφυλακής. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή Αλίας δεν έχουμε κανέναν. Οπότε θα δώσω το λόγο σε δύο συναδέλφους αν συμφωνείτε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των τριών οργανισμών για την εκτενή παρουσίαση. Έδειξαν τις συνέργειες που υπάρχουν. Επανέρχομαι στην αρχική δήλωση, γιατί πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο έγινε μετά από τις εικόνες που είδαμε το 2015. Και σύντομα ήθελα να πω ότι οι εικόνες του 2015 δημιουργήθηκαν επειδή τα κράτη-μέλη και οι οργανισμοί δεν κόπιασαν να βρουν ε, τρόπους αντιμετώπισης των αιτίων της φυγής και δεν αντιμετώπισαν τον αριθμό των μεταναστών που έρχονταν στην Ευρώπη με τρόπο επαρκή. Έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση προς τους εκπροσώπους των τριών οργανισμών. Αν μπορούμε να εντοπίσουμε τα σκάφη που κινούνται στη Μεσόγειο, να δούμε δηλαδή το δρομολόγιο που ακολουθούν, τι θα γίνει. Αν ας πούμε η ΕΜΦΚΑ δει ένα σκάφος με μετανάστες ή πρόσφυγες, μετά τι θα γίνει. Δεύτερον, αν διαπιστώσετε ότι ένα γερμανικό πλοίο με πρόσφυγες φύγει από τις λιβικές ακτές, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Και τρίτον, οι ακτές της Λιβύης παρακολουθούνται εντονότερα ενώπιση των εξελίξεων ε, και καταγράφονται τα πλοία που φεύγουν με πρόσφυγες μετανάστες από εκεί. Θα έπρεπε να έχουμε πιο πολύ χρόνο για τη συζήτηση και δυστυχώς δεν έχουμε για να τα αναπτύξουμε όλα αυτά. Λοιπόν, κυρία Γκρίσμπα, και μετά θα δώσουμε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ τους εκτελεστικούς διευθυντές των οργανισμών που μας παρουσίασαν ε, την ε, έκθεση αυτή. Είναι Δευτέρα, ξεκινάει η εβδομάδα, δεν είχαν φτάσει όλοι οι συνάδελφοι, αλλά θα διαβάσουν τα πρακτικά οι συνάδελφοι. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν όσον αφορά την κοινή χρήση των μέσων και τον επιμερισμό των διαδικασιών ε, και κυρίως ε, των ε, επιχειρήσεων ε, στην θάλασσα, όχι τόσο στις, ε, σε χερσαία σύνορα και στις ακτές. Ε, λυπούμε όμως που μια τέτοια δραστηριότητα δεν, είναι, δεν, γίνεται γνωστή στους πολίτες. Γίνονται τόσα πράγματα όσον αφορά και την παράτιμη μετανάστευση και όσον, τη διάσωση των ανθρωπίνων ζώων, όσον αφορά το και όσον αφορά τις εγκληματικές δραστηριότητες κτλ. Και ο κόσμος δεν το ξέρει, οι πολίτες δεν το ξέρουν διάσωση ε, στη θάλασσα βεβαίως ε, ε, παίρνει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις, σοβαρές διαστάσεις σε όλο τον κόσμο. Ε, πρέπει να πούμε ότι και ε, ε, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ειρηνικό ωκεανό, κυρίως όσον αφορά ε, ζώνες αποκλειστικής αρμοδιότητας γύρω από, την νήσο της Ρεϊνιό, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και όσον αφορά αλληλεία, παράνομες αλληλευτικές δραστηριότητες κτλ. Και επίσης όσον αφορά την διάσωση ανάμεσα στις νήσους Κομόρες και την Μαγιότ έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που χάνουν ε, την ε, ζωή τους ε, προσπαθώντας να φτάσουν σε αυτό το Ελντοράντο που πιστεύουν ότι είναι το, το, το νησί της Μαγιότ. Η κατάρτιση είναι πολύ σημαντική, την αναφέρατε. Εγώ και το είδος των αποστολών επίσης και των επιχειρήσεων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 67 εκατομμύρια ευρώ ε, για, το, για, το, για την υπηρεσία αυτή. Ε, στις παρουσιάσεις σας αναφερθήκατε και στην χρήση μη επαδρομένων αεροσκαφών, ντρόν ε, κτλ. Όμως, να ρωτήσω το εξής. Ε, αυτό το σύστημα ε, των τηλεκατευθυνωμένων ε, αεροσκαφών εκτός από τα drones αναπτύσσεται παράλληλα ε, ε, έπρεπε να είναι λειτουργικό πλήρω τον Ιούνιο του 2017. Τι γίνεται με αυτό. Ε, επίσης, μια και πρόκειται για πιλωτικό πρόγραμμα, περιμένουμε βεβαίω και αποτελέσματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, συγκεκριμένα στοιχεία. Και τέλος, ποιο θα είναι το μέλλον της διαδικασίας. Θα εξακολουθήσετε, όπω και εγώ το εύχομαι, αυτέ τι κοινέ επιχειρήσει και δραστηριότητε ή θα σταματήσουμε κάποια στιγμή και δεν θα κάνουμε, δεν θα συνεχίσουμε ε, με κάτι με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους τρεις εκτελεστικούς διευθυντές ε, που προσήλθατε στη σημερινή μας ε, συνεδρίαση καθώς πρόκειται για ένα περίπλοκο τομέα συνεργασίας. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κι εγώ ένα ερώτημα από τη δική μου πλευρά. Λίγο πριν από τη σημερινή συνεδρίαση είχαμε κάνει μια συζήτηση μεταξύ των συντονιστών και το πρώτο ερώτημα που είχε τεθεί ε, βέβαια ε, ήταν ακριβώς αυτό ως το τι συμβαίνει με την υπηρεσία ε, συνοριοφυλακής. δημιουργείται πώς, πώς πάμε, ποια είναι η πρόοδος. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς γίνεται η διαχείριση, γιατί έχετε μια σειρά από τομείς δραστηριότητες, μόλυνση, αλληλεία, μεταφορές ε, και βέβαια κυρίω ε, έχουμε να κάνουμε την αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την διαχείριση των συνόρων και τη μετανάστευση. Άρα λοιπόν πώ διαχειρίζεται τι προσδοκίε ε, όλων αυτών που αναμένουν πολλά να επιτευχθούν στο πλαίσιο τη συνοριακή και ακτοφυλακή μέσα στα επόμενα χρόνια. Γνωρίζετε πω υπάρχουν αυτέ οι προσδοκίε από την πλευρά των κρατομελών ή προσπαθείτε να δώσετε περισσότερη έμφαση σε μια συνεργατικό αν θέλετε χαρακτήρα σχέση με τα κράτη-μέλη. Τι είδου δηλαδή εταιρική σχέση δημιουργείται με τα κράτη-μέλη. Οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια ο καθένα από τη δύο πλευρά, λαμβάνοντα στο βαθμό που μπορείτε υπόψη τα σχόλια και τα ερωτήματα που έκαναν οι συνάδελφοι. Ποιο θέλει να ξεκινήσει, ο κύριο Μούλη. Μπορείτε θέλετε να επανέλθετε με την σειρά που κάνετε για τι παρουσιάσει σα, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ όσου έθεσαν αυτά τα ερωτήματα. Ναι, πράγματι, Φανταζόμαστε ότι υπάρχουν ε, μεγάλες προσδοκίες από τα κράτη-μέλη και από τους νοικόμενους ε, ε, φορείς σε ό,τι αφορά αυτήν την ακτοφυλακής γιατί βέβαια αποτελεί και μια πρόκληση για τα κράτη-μέλη, αλλά και τελικά για τους συμμετέχοντες στα διοικητικά συμβούλια αυτών των τριών οργανισμών ως προς το πώς θα λειτουργήσει. οι τρεις οργανισμοί μας έχουν δημιουργήσει μια συμφωνία, αν θέλετε, λειτουργίες ε, τρίμερη, working arrangement, όπου έχουμε ορίσει ακριβώς τα καθήκοντα και τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ μας. Επίσης έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από τεχνικού χαρακτήρα υποομάδες, από διαφορετικές υπηρεσίες, οι οποίες προωθούν ουσιαστικά τη συνεργασία μας περισσότερο σε μια σειρά από διαφορετικούς τομείς. Άρα λοιπόν θέλουμε να τονίσουμε ότι ο κάθε οργανισμός ε, απευθύνεται σε, μια, σε, σε, διαφορετικούς, σε διαφορετικές ομάδες στόχους, σε διαφορετικούς φορείς, στα κράτη-μέλη, που στα, ε, στο πεδίο αρμοδιότητας του καθενός από αυτούς. Άρα λοιπόν αυτό που ε, θέλουμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε περισσότερο τους πόρους μας, να αξιοποιήσουμε περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας, αλλά χωρίς να παρεκκλίνουμε από τις ομάδες στόχους μας, από, δηλαδή τους φορείς τους οποίους προσφέρουμε τα όσα προσφέρουμε. Είναι γεγονός ότι έχουμε ε, δημιουργήσει μία εκτελεστική επιτροπή, implementing group, κυρίως για τη Μεσόγειο όπου για τις επιχειρησιακές ε, διαδικασίες οι εμπειρογνώμονες ε, των ε, κρατών μελών που προέρχονται από τον τομέα του ελέγχου της Ελίας και από τον τομέα του ελέγχου των συνόρων συνεργάζονται και συναντώνται τακτικά. Ξεκίνησε αυτό την αρχή του 2016 τότε που ξεκίνησε και η συνεργασία ε, με την ε, Frontex και ε, αυτή η πλευρά είναι ιδιαίτερως αποτελεσματική. Thank very much. Uh, Mr. if you conclude, please. Και εσείς παρακαλώ για να ολοκληρώσετε. Να πω... Σε, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες διάσωσης να σας πω το εξής. Μα από αφορά της Frontex, όταν εμείς διαπιστώσουμε, διαπιστώνουμε ότι ένα πλοίο αναχωρεί από τη Λιβική Ακτή με μετανάστες, αυτό μπορούμε να κάνουμε να διαβιβάσουμε αυτές τις πληροφορίες στα κράτη-μέλη. Αλλά η ίδια υπηρεσία, ο ίδιος ο δεν μπορεί ε, δεν έχει κάποιο σημείο επαφή στη Λιβύη, οπότε δεν μπορεί να αναλάβει δράση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαβάσουμε αυτή την πληροφορία στα κράτη-μέλη. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια ω προ τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού έργου. Ε, Προφανώ πρόκειται για μια πολύ επιτυχή συνεργασία μεταξύ των τριών οργανισμών, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων, αν θέλετε, φορέων δηλαδή, ε, με αρμοδιότητε Ε, ε, σε ό,τι αφορά τις πτυχές της φύλαξης των συνόρων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με ε, περισσότερο αποτέλεσμα που μπορούμε να επιτύχουμε σε ό,τι αφορά την επιβολή της νομοθεσίας στη θάλασσα. Δηλαδή, όταν προσπαθούμε για παράδειγμα να καταπολεμήσουμε και το διασυναριακό έγκλημα, έχουμε εδώ ακριβώς ένα συμπληρωματικό πλεονέκτημα, για παράδειγμα στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ΕΜΣΑ, γιατί μπορούμε να διαπιστώσουμε, για παράδειγμα, εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ε, ε, για παράδειγμα επιθεωρήσεων σε ό,τι αφορά την παράνομη αλληλεία. Αυτές λοιπόν οι πληροφορίες μπορούν να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε με τις τελωνιακές αρχές των κρατών μελών, αλλά και στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας ε, που έχουμε για παράδειγμα μεταξύ Frontex και Europe. Οπότε κατά τη δική μου άποψη πρόκειται εδώ για ένα υβριδικού χαρακτήρα αν θέλετε έργο το οποίο μας καταδεικνύει το τι θα μπορούσε να προκύψει ω μέθοδο συνεργασία μεταξύ αυτών των οργανισμών και των ε, υπηρεσιών των κρατών μελών. Ένα είδο δηλαδή δημόσια υπηρεσία, αν θέλετε, όπου ο καθένα, ο κάθε συμμετέχοντα, ε, σέβεται πλήρω την εντολή και τα καθήκοντα του κάθε συμμετέχοντα φορέα και του κάθε συμμετέχοντα οργανισμού, αλλά ταυτόχρονα όλοι οι συμμετέχοντε ε, προσφέρουν και διαχειρίζονται από κοινού τι δυνατότητε του, τι ικανότητες του και μοιράζονται τι πληροφορίε του. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, αν θέλουμε να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε δρόση όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, όταν υπάρχει για παράδειγμα ζήτημα σύλληψη ε, διακινητών ελαφρομεταναστών, εάν πρόκειται για ένα ζήτημα διάσωση, εάν πρόκειται για ένα ε, ε, ζήτημα περιβαλλοντική διάσωση, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε δράση. Άρα λοιπόν διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες αλλά και διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τις ικανότητες. Είναι σημαντικά λοιπόν αυτά τα στοιχεία και ε, το πιλωτικό έργο θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε ένα είδος κοινών προτύπων, δηλαδή τυποποιημένων διαδικασιών που θα, που θα ακολουθούμε αλλά και τεχνικά πρότυπα που θα εφαρμόζουμε. Μέσα στους επόμενους ε, μήνες ε, θα υπάρξουν συναντήσεις ε, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ακτοφυλακής και επίσης θα υπάρξουν και περισσότερες επαφές σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν βέβαια και περιοχές σε περιφερειακό επίπεδο που θα μπορούσαμε να ε, προβούμε σε μια πιο συγκεκριμένη συνεργασία. Αυτά από την πλευρά μου και θα ήθελα για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εμπιστοσύνη που μα επέδειξαν ε, και την οποία εξέφρασα σήμερα εδώ από την πλευρά και των τριών επιτροπών. Ευχαριστώ λοιπόν και την ε, Επιτροπή για την υποστήριξή τη και για τα κράτη-μέλη αλλά και τον Πασχάλ και τον Μάκο και τι ομάδε από, τους, από την πλευρά των τριών οργανισμών για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε μεταξύ μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό θα ήταν να ε, υπάρχει δυνατότητα πιο συχνών συναντήσεων όπως αυτή. Ευχαριστώ όλους ε, τους τρεις εκτελεστικούς διευθυντές. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία και βεβαίως δείξατε και τις προκλήσεις και τα επόμενα βήματα και εμείς ε, και οι συγητές και τα ενδιαφερόμενα μέλη θα παρακολουθούμε προσεκτικά τους φακέλους. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή ε, Μεταφορών για την παρουσία της εδώ, τις παρεμβάσεις της. Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσουμε την επαφή μας σε λίγους μήνες να δούμε πώς συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Uh, λοιπόν, να προχωρήσουμε γρήγορα στο επόμενο σημείο, το 5, για τις συμφωνίες επανεισδοχής. If to come to the for the Okay, um, Συνάδελφοι, αν είστε έτοιμοι και επειδή περνάει ο χρόνος πολύ γρήγορα, ας πάμε στο επόμενο θέμα. Τώρα θα κάνουμε μια, την κανονική αξιολόγηση από την πλευρά της Επιτροπής μας σχετικά με την κατάσταση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες επανεισδοχής. Έχουμε προσκεκλημένο για μια παρουσίαση, θα πω κι εγώ δύο λόγια όμως σχετικά. Ο Σάιμον, ο κύριος Μορντιού, ήρθε στις 7 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα θυμάστε όταν κάναμε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και την υλοποίηση των συμφωνιών επανεισδοχής γενικά. Ξέρετε ότι απίφθηνε επιστολή στον Επίτροπο πριν από λίγες εβδομάδες και είπε ότι ανησυχούμε για την αυξημένη χρήση άλλων μέσων που δεν έχουν την νομοθετική μορφή συνεργασίας με τρίτες χώρες για την επιστροφή επαναπατρισμό των ε, πολιτών τους που είναι παράνομοι εδώ. Επίσης ε, αναφέρθηκα στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση που αναφέρει ότι παράλληλα με τις επίσημες διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει και άτυπες ρυθμίσεις. Επέστησα την προσοχή του Επιτρόπου στο γεγονός ότι οι άτυπες ρυθμίσεις με τρίτες χώρες για την επανεισδοχή ε, απασχολούν ιδιαίτερα την Επιτροπή γιατί το Κοινοβούλιο μπορεί να μην μπορεί να ε, αποφαίνεται όπως προβλέπει το άρθρο 218 της Συμφωνίας για τη Λειτουργία την ε, για τη Συμφωνία για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συζητήσαμε για, ήδη για πολλά ενδιαφέροντα θέματα και χαίρομαι που ο Σάιμον επανήλθε έγκαιρα για να μας ενημερώσει. Ε, αυτή είναι ε, δημόσια συνάντηση, θυμίζω. Τώρα Χωρίς ε, άλλη καθυστέρηση δίνω το λόγο στον Σάιμον. Κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητά μέλη, ε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε επαναπατρισμό αυτών που δεν δικαιούνται να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η επανεισδοχή από την χώρα τους. Θέλω να καλωσορίσω και εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια Τινησίας και Μαρόκο που είναι οι εταίροι μας στη διευθέτηση του μεταναστευτικού. Ε, σίγουρα θα πρέπει να τονίσουμε το σεβασμό προς, τα, προς κάθε άνθρωπο και θα πρέπει να προβλέψουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη προστασία. Θα ήθελα λοιπόν να πω για την ευρύτερη στρατηγική μας μερικά πράγματα, τονίζοντας ότι η επιστροφή και η επανεισδοχή δεν είναι η αποκλειστική μας στόχη. Ο στόχος μας είναι ένα πλαίσιο προβλέψιμο που θα βρει σωστή ισορροπία μεταξύ ελληνικής υπευθυνότητας, αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς ε, κρατούμε ανοιχτά τα ενδεχόμενα και δυνατότητε προστασίας για αυτού τους ανθρώπους. τι προκλήσεις θέλουμε να τι αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αλλά και με τρόπο ανθρώπινο. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση δηλαδή ε, για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, για τις ε, οδούς προς την Ευρώπη, και δουλεύουμε με βάση εταιρικέ σχέσεις εντός και εκτός της Ένωσης. Ακούσατε τον Φαμπρίς, εργαζόμεθα και με χώρες εταίρους για να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα. Ε, δουλεύουμε για να αντιμετωπίσουμε τα αίτια και τις ρίζες του μεταναστευτικού ε, για την προστασία των μεταναστών και την καταπολέμηση των διακινητών, των λανθρεμόρων. Και είχαμε κάποια αποτελέσματα ήδη σε πολλούς τομείς εργασιών μας. Συνεργαζόμεθα επίσης και με τον IOM και την UNHCR. Ε, ε, Η Λιβύα ήταν στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες Τονίζω ότι περίπου 4.000 μετανάστες και πάνω από 2.000 εκτοπισμένες οικογένειες ε, πήραν ε, στήριξη ε, και ιατρική βοήθεια μεταξύ άλλων. Βεβαίως θέλουμε να βάλουμε τέλος στα αυτά τα φρικτά κέντρα κράτησής τους. Δεκάδες χιλιάδες ε, ε, άνθρωποι από την Λιβύη μεταξύ άλλων ωφελήθηκαν από τη δυνατότητα ε, επαναπατρισμού. Υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του αριθμού. Είδαμε και κάποια παραδείγματα mm. περιορισμένου αριθμού ανθρώπων που πήγαν από τη Λιβύη στην Ισία και τώρα θέλουμε να, ε, σε εκούσια βάση ε, να επιστρέψουν. Εξετάζομαι τα αίτια του κακού, χρηματοδοτούνται προγράμματα για το, μέσα από το Trust Fund τη, για την Αφρική θέλουμε να στηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη, τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Υπάρχουν ιδιωτικέ επενδύσει 14 ε, εκατομμυρίων ευρώ που είναι τώρα στη διάθεσή μα ε, και στην ε, επανεγκατάσταση προχωρήσαμε καλά. Τώρα έχουμε 34.000 θέσεις μετεγκατάστασης και αυτό δείχνει τη δέσμευση των κρατών μελών να μειώσουν την ε, επικίνδυνη έλευση των ε, μεταναστών. Τα λέω αυτά ε, ευθύ εξ αρχής γιατί αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι το έργο της Κομισιόν δεν θέλει να κάνει φρούριο την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλα αυτά τα μέτρα προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι θα μείνουμε ένα ασφαλές λιμάνι για αυτούς που χρήζουν προστασίας. Αλλά νομίζω ότι για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα ε, το επίπεδό μας και να δώσουμε προστασία σε αυτούς που τη χρειάζονται, ε, θα πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Ε, να δούμε δηλαδή εκείνους που δεν μπορούν να παραμείνουν στην Ένωση μετά από σωστή εξέταση της περίπτωσης. Εκείνοι που δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν λοιπόν θα πρέπει να επιστρέψουν. Και έτσι περνώ στο σημερινό μου θέμα, δηλαδή τις προκλήσεις επαναπατρισμού και επανεισδοχής. Παραμένει μεγάλη πρόκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αν δείτε τα πρόσφατα στοιχεία, ε, περίπου 36% των παράτυπων μεταναστών μετά από ε, εξατομικευμένη διαδικασία ε, ασύλου επιστρέφουν. Και υπάρχουν πολλές προκλήσεις σε σχέση με τα εθνικά συστήματα επιστροφών στα κράτη-μέλη. Ε, κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε τη συζήτηση της επόμενης εβδομάδας που θα επικεντρωθεί σε αυτά τα θέματα. Ως Κομισιόν στηρίζομαι τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές τους να ξεπεράσουν αυτά τα εσωτερικά εμπόδια στην ε, αποτελεσματική επιστροφή. Η, εκούσια επιστροφή ε, παραμένει η προτιμόμενη λύση για την Κομισιόν και την Ένωση. Εμείς παρέχουμε σημαντική οικονομική βοήθεια στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να γυρίσουν στα πλαίσια ενός ε, εκούσιου συστήματος. Υπάρχουν ε, πακέτα επανένταξή τους για αυτό το σκοπό. Αν δούμε κάποια δεδομένα που δίνουν τα κράτη-μέλη και τα έχετε λάβει πριν από την συνάντηση αυτή, γιατί είναι πολλά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιστροφές. Ελπίζω να καλύψαμε έτσι το αίτημα που διατυπώσατε ως Επιτροπή την προηγούμενη φορά, που θέλατε στοιχεία για τις επιστροφές και επίση, αν θέλετε και άλλε πληροφορίε για αυτό το θέμα ή για οποιοδήποτε άλλο θα σα δώσουμε αργότερα. Και βλέπετε με βάση τα νούμερα λοιπόν υπάρχει μια μικρή αύξηση στον αριθμό των οικουσίων επιστροφών από 39.000 το 2015 στι 46.000 το 2016. Και εδώ θα έλεγα όμω ότι ένα λόγο που είδαμε αυτή την αύξηση των οικουσίων επιστροφών είναι ότι η προοπτική τη αναγκαστική επιστροφής ακούσια ενθαρρύνει τον κόσμο να επιλέξει την εκούσια επιστροφή. Επίσης η εκούσια επιστροφή σε πολλές περιπτώσεις είναι πιθανή αν δεν ε, υπάρχει και η προοπτική της αναγκαστικής επιστροφής και έτσι περνάω στην καρδιά του προβλήματος. Νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι τα κράτη-μέλη συχνά ακόμα αντιμετωπίζουν έλλειψη συνεργασίας από τις χώρες προέλευσης και τις αρμόδιες αρχές εκεί. Παράδειγμα, όταν κάποιος δεν έχει έγκυρο διαβατήριο και επιστρέφει, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απευθυνθούν στο προξενείο της χώρας για να δώσουν ένα ε, ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο πολλές φορές θα χρειαστεί και συνέντευξη για αυτό το πράγμα. Για αυτά τα δύο βήματα χρειάζεται συνεργασία με τις χώρες εταίρους. Και συχνά είναι δυσχερής αυτή η συνεργασία. Κάποια προξενία δεν ταυτοποιούν τους ε, υπηκόους τους αν θεωρούν ότι ε, υπάρχει το ενδεχόμενο της αναγκαστικής επιστροφής. Και αυτό δεν δείχνει μόνο ε, μη σεβασμό στο δικαίωμα του κράτου, με, κράτους μέλους να αποφασίσει ποιος θα μπει στο, και θα μείνει στο έδαφος του, αλλά καμιά φορά αμφισβητεί και την υποχρέωση των χωρών εταίρων στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου να πάρουν πίσω τους ε, υπηκόους τους. Η, η ε, επανεισδοχή είναι υποχρέωση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και όταν μιλάμε με τους εταίρους από την υποσαχάρια περιοχή είναι και υποχρέωση με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Συμφωνία του Κοτονού και το άρθρο 13 που προβλέπει πολύ ισχυρή νομική βάση και είναι και πολλές φορές αυτοδικαίωση για τις χώρες και μια συμφωνία επανεισδοχής. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν πολλές φορές είναι πρακτική ρύθμιση ώστε αυτές οι επανεισδοχές να γίνουν στην πράξη. Ε, αυτό εν μέρει εξηγεί γιατί συχνά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νομικά μη δεσμευτικές ρυθμίσεις επανεισδοχής που ε, πρόκειται να θέσουν σε εφαρμογή τις νομικές υποχρεώσεις που υπάρχουν στο άρθρο 13 του Κοτονού. Ε, αυτές δεν είναι νομι, νομι, νομικές υποχρεώσεις, αλλά ε, ε, ρυθμίσεις ε, που θα λάβουν υπόψη τις διεθνείς ρυθμίσεις για να πραγματοποιηθούν οι επανεισδοχές. Και το αποτέλεσμα αυτών των ρυθμίσεων μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Επίσης, να σας πω ότι η προτιμόμενη επιλογή για την Κομισιόν είναι πάντοτε όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις που υπάρχουν και που θα ενδυναμώνονται μέσα από συγκεκριμένες συμφωνίες επανεισδοχής. Αλλά αυτό δεν γίνεται πάντοτε, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά που ήρθα, με κάποιες χώρες εταίρους ε, και με δεδομένες τις πολιτικές ευαισθησίες της χώρας ε, καταγωγής. Όταν οι τρίτε χώρε είναι απρόθυμες λοιπόν να συνάψουν συμφωνίε επανεισδοχή, θα πρέπει από την πλευρά μα να δείξουμε κάποια ε, ευελιξία, ε, να είμαστε επικοδομητικοί και να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα πάντα στα πλαίσια της, του σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Ε, το 2017 είχαμε κάποια αποτελέσματα. Να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες τώρα σε σχέση με την πρόοδο αναχώρα και με τις χώρες με τις οποίες συνήψαμε ε, διοικητικές ρυθμίσεις ε, και αυτές που έχουν πιο επίσημες ε, συμφωνίες επανειδοχής. Τις δύο χώρες καταρχήν που αναφέρονται στον τίτλο της παρουσίασης, το Μάλι και το Αφγανιστάν. Αρχίζω με το Μάλι. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για τις πολιτικές ευαισθησίες και για τη διακριτική ευχέρεια που πρέπει να δείχνει η Ένεση πολλές φορές. Το Μάλι αποσύρθηκε από την ολοκλήρωση των ε, των ε, τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών ε, σχετικά ε, όταν έπρεπε να υπογραφεί η επίσημη συμφωνία. από, τόνισαν ότι ε, δεν ε, ε, υπέγραψαν επίσημη συμφωνία, δεν έλαβε χώρα κάτι τέτοιο. Οι αρχές του Μάλι εργάζονται καλά όμως με μας, διευκολύνοντας την εκούσια επιστροφή των υπηκόντους που είναι στη Δυνησία και στη Λιβύη. Όμως ε, δεν έγινε πρόοδος για να βρεθεί τρόπος ε, ε, επίσημης επανεισδοχής μετά από τα περσινά εμπόδια. Οπότε δεν υπάρχει συμφωνία επανεισδοχής ούτε ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή με το Μάλι. Για το Αφγανιστάν η υλοποίηση του Joint Way Forward, κοινό τρόπος για να πάμε μπροστά, αυτό συνεχίζεται από τότε που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2016 περίπου 19 πτήσεις charter έγιναν με περιορισμένο αριθμό, δηλαδή 287 επαναπατριζόμενους. Θα συνόψιζα την ικανοποίηση των κρατών μελών λέγοντας ότι γενικά είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τις αφγανικές αρχές και βρέθηκε μια καλή πλατφόρμα για να συζητηθούν πιθανά εμπόδια στη συνεργασία. Αυτή η προοπτική της αναγκαστικής επιστροφής σε περιορισμένες περιπτώσεις ήταν ένας παράγων για τους οποίους ο ολικός αριθμός των επιστροφών αυξήθηκε από 1.500 επιστροφές το 2015 στις 8.325 το 2016. Είδαμε επίσης πολύ σημαντική πτώση στις αφήξεις των παράνομων μεταναστών από το Αφγανιστάν από 54.000 το 2016, τώρα έχουμε περίπου 4.000 από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτό έπαιξε ρόλο. Τώρα το Μπαγκλαντές, εκεί ε, ε, είχαμε πάρα, πολλούς, πάρα πολλές αφήξεις, 9.000 ε, αφήξεις από τις αρχές του 2017. Το Σεπτέμβριο ε, από την πλευρά της Κομισιόν και της Ένωσης συμφωνήσαμε με τον Μπαγκλαντές για ε, τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες ε, ώστε να επιστρέψουν ε, οι υπήκοοι του Μπαγκλαντές όταν δεν δικαιούνται άσυλο και δεν έχουν λόγο να μείνουν. Τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους θα δώσω στοιχεία. Η Ουγγνία είναι μια χώρα 12 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ε, ε, μέσα από την Κεντρική Μεσόγειο ε, έρχονταν πάρα πολλοί μετα, ε, μετανάστες. Η συνεργασία ήταν φτωχή. 5% ήταν το ποσοστό επιστροφών, αλλά τον Ιούλιο φέτος μπορέσαμε να κάνουμε συμφωνία ορθών πρακτικών για την αποτελεσματική ε, οργάνωση της διαδικασίας επιστροφής και οι πρώτοι ε, παναπατριζόμενοι έφυγαν. Θα αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, γιατί βλέπουμε ότι πηγαίνει καλά αυτό. Αιθιοπία, θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία για την ταυτοποίηση με την Αιθιοπία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και συχνά η Αιθιοπία αρνεί να ε, δεχτεί τους υπηκόους της, εκτός και αν συμφωνούσαν να επιστρέψουν. Τους τελευταίους μήνες δίναμε ε, τη συνεργασία και τώρα σκεφτόμεθα να εισαγάγουμε ορθές πρακτικές για την επιστροφή, ώστε να κάνουμε κάποια πρόοδο. Αυτά είναι υποσυζήτηση τώρα με την Αιθιοπία. Ε, άλλες χώρες από την Αφρική ακτή του Ελεφαντοστού που είναι η τρίτη χώρα προέλευσης παράνομων μεταναστών. Το ποσοστό επιστροφής ε, στη χώρα αυτή, όπως ε, είδατε από τα στοιχεία, είναι χαμηλό, περίπου 5%. Feedback δεν έχουμε λάβει ακόμα από την ακτή του ελεφαντοστού, δηλαδή προτάσεις για να βρεθούν, ρυθμίσεις για να βελτιωθούν ε, και να αυξηθούν οι επιστροφές και με την Γκάνα επίσης θέλουμε συνεργασία γιατί είδαμε μια σταθερή αύξηση παράνομων αφήξεων τα τελευταία χρόνια από την Γκάνα. Και εδώ προτείνουμε να βρούμε πρακτικές ρυθμίσεις που θα σέβονται τις ευαισθησίες των εταίρων. Ακόμα όμως περιμένουμε την απάντηση από την Γκάνα. Επίσης, μετά την δημοκρατική αλλαγή στην Γκάμπια και τη θετική αυτή αλλαγή, Κάναμε συζητήσεις με τη χώρα αυτή για να βρεθούν παρόμοιες ρυθμίσεις. Αυτά για τις χώρες ΑΚΕ, όπου έχουμε και ισχύει το άρθρο 13 της Συμφωνίας του Κοτονού και παρέχει νομική βάση. Τώρα πολύ γρήγορα επανέρχομαι στους τομείς όπου έχουμε επίσημες συμφωνίες ε, ε, πανισδοχής. Να σας ενημερώσω σχετικά με το τι έγινε μετά τις 7 ε, Σεπτεμβρίου. Ας δούμε το Πακιστάν. Το Σεπτέμβριο είχαμε ε, μια κοινή επιτροπή επιστροφών με το Πακιστάν και μπορέσαμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση με το Υπουργείο Εσωτερικών ιδιαίτερα για την ανάγκη να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ε, ε, και να ε, επιστρέψουν οι άνθρωποι που είχαν ε, φτάσει στην Ελλάδα μεταξύ άλλων. Εδώ δημιουργούμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών που θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις αιτήσει επανεισδοχής. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο θα τρέξει δοκιμαστικά Τώρα, οι χώρε ε, Δυτικών Βαλκανίων και Ανατολικής ε, σχέσης γειτονία, εδώ έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά επιστροφών, 84% στην Ουκρανία, ε, κάποιες δυτικές, χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουμε παρόμοια ποσοστά που καμιά φορά υπερβαίνουν και το 100%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε επιστροφές από την καθυστέρηση που υπήρχε από τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο για τη ΦΥΡΟΜ. Γενικά λοιπόν θα έλεγα ότι η συνεργασία με τις χώρες ε, των Δυτικών Βαλκανίων είναι υποδειγματική στον τομέα των ε, παναπετρισμών. Το ίδιο και με τη Μολδαβία. Πολύ γρήγορα για την Τινησία, επίκαιρο θέμα αφού έχουμε και φίλους από την Τινησία εδώ. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Αν δούμε τα στοιχεία των αφήξεων στην Ιταλία, μόνο για τον Οκτώβριο η Τινήση ήταν περίπου 2.788, ε, ε, περίπου το 50% όλων των αφήξεων τον Οκτώβριο στην Ιταλία. Έχουμε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Τινησία που προγραμματίζεται στις 28 Νοεμβρίου να δούμε δηλαδή συμφωνίες διευκόλυνσης θεωρήσεων και μια συμφωνία πανεισδοχής ένωσης Ισία. Θα ενημερωθείτε, θα φροντίσω άμεσα να ενημερωθείτε. Διαπραγματεύσεις γίνονται και με την Ιγυρία. Οι διαπραγματεύσεις αυτές άρχισαν τον Οκτώβριο του 2016 και ακόμα όμως ε, ε, είναι στάσιμες. Ε, θα ήθελα τέλος ε, να πω ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, οι προκλήσεις ε, επιμένουν, ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα συμφέροντα αυτών των προσώπων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επίσημε συμφωνίε επανεισδοχή. Η συνεργασία σε και η εταιρική σχέση ε, είναι η προσέγγιση μα και από την πλευρά τη Ένωση θα πρέπει να σκεφτούμε πώ μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε κίνητρα εξατομικευμένα, να τα προσφέρουμε στους ανθρώπου αυτούς, ώστε οι εταίροι μα να θέλουν να συνεργαστούν μαζί μα. Μην ξεχνάμε και το σεβασμό που οφείλουμε στις ευαισθησίες αυτών των χωρών εταίρων, ιδιαίτερα ε, επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της έλλειψης ικανοτήτων ε, για να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση. Τέλος, ο, εάν θέλετε οποιασδήποτε λεπτομέρειες για τις ε, διευθετήσεις αυτές, τις διαπραγματεύσεις που διεξάγουμε, θα σας στείλουμε στοιχεία ε, ευχαρίστως ε, σημαντικές λεπτομέρειες αν θέλετε να λάβετε υπόψη σας ε, κάποια λεπτά ζητήματα που αφορούν επιμέρους χώρες. Ευχαριστώ. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου της Εθνικής και του Μαρού και θα δώσω κάποια στιγμή τη δυνατότητα και σε κάποιους εκπροσώπους τους να πάρουν το λόγο αφού πάρουν τα μέλη ε, το λόγο τα μέλη εδώ τη Επιτροπή ΕΛΙΒΕ. Του ευχαριστώ πάντω ε, για την ε, παρουσία του σήμερα εδώ, ειδικότερα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Αφρική. Τώρα, να σα διαβάσω ποιοι θα είναι οι ομιλητέ μα για αυτό το σημαντικό ζήτημα, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν ότι πράγματι έχουν περιληφθεί εδώ στον κατάλογο των ομιλητών. Όλμαρ, Κιέγκε, Τεβέα, Σαρτζεντίνη, Γιόρκ, την Κρεπίνη. Αν Κριστίν θέλεις να πάρεις και εσύ το λόγο. Είσαι σίγουρο ότι θέλεις να πάρεις το λόγο και εσύ. Καλώς. Γιατί βέβαια θα χρειαστεί να ακάσουμε και σε απαντήσει από πλευρά του κ. Μωρίδη. Οπότε ας ξεκινήσουμε με την κυρία Ρουμαρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω κύριο Μορντού για αυτήν την ε, εις βάθος παρουσίαση ε, και την ε, ράση αν θέλετε εδώ που μας παρουσίασε των άτυπων αν θέλετε διακανονισμών με χώρες με τις οποίες δεν έχουμε κάποια επίσημη συμφωνία και αυτός ο αριθμός των 34.000 σε ό,τι αφορά τις, το resettlement την εσωτερική μετακατάσταση είναι ενθαρρυντικός όπως όλοι γνωρίζουμε ε, μία οργανωμένη πολιτική επιστροφών συμβάλλει ε, σε αυτό και ε, θα ήθελα να ζητήσω μια διευκρίνηση συμβάλλει δηλαδή και στο να ενθαρρυνθούν περισσότερο οι εθελούσιες επιστροφές και ότι δηλαδή είναι δυνατόν να ληφθούν περισσότερα μέτρα και να προωθηθούν αυτέ και συνοδευτικά μέτρα σε ό,τι αφορά αυτέ τι θελούσε επιστροφέ. Ε, θα ήθελα να, να μα πείτε και ε, λίγε παραπάνω λεπτομέρειε σε ό,τι αφορά τι θελούσε επιστροφέ, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα πρόβλημα που έχουμε βιώσει σε ό,τι αφορά τι επιστροφέ στη δική μα χώρα. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία έχουν ε, εισέλθει παρατύπωσε στη δική μας επικρατεία και από τα οποία ε, ζητείτε να επιστρέψουν στις χώρες τους τα προσεγγίζουν πολύ στοχευμένα ε, δίκτυα ε, πρόθεσης λαθρομετανάστευσης και τα οποία ε, προσπαθούν να αξιοποιήσουν την, την, την, την κατάστασή τους έτσι ώστε να εξαφανιστούν αν θέλετε από το ραντάρ. Γνωρίζοντας δηλαδή ότι από τη μία πλευρά επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, από την άλλη όμως δεν το επιθυμούν και έτσι ε, αυτό που κάνουν αυτά τα δίκτυα ελατρομετανάστευση είναι να προσπαθούν να στρατολογήσουν εντό εισαγωγικών αυτά τα άτομα για συγκεκριμένε εγκληματικέ ε, δραστηριότητε. Ουσιαστικά δηλαδή να τα εκμεταλλευτούν προκειμένου να ε, συμμετάσχουν. Οπότε έχετε εσεί προβλέψει κάποια μέτρα έτσι ώστε να αποτρέπεται καταρχήν αυτή η εξαφάνιση εντό εισαγωγικών των ατόμων από τα οποία συζητηθεί να αποχωρήσουν ε, και πώ επίση, αν ε, υπάρχουν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η στρατολόγηση αυτών των ατόμων για κλιματικέ δραστηριότητε. Ευχαριστώ, πρόεδρο. ο Πρόεδρο. Ε, σα παρακαλώ όλοι να περιορίσετε σε δύο λεπτά στι παρεμβάσει σα. Κύριε Γκέγκε, το έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν συμμερίζομαι ε, την λογική του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Κυρίως όταν τα μέσα ε, είναι συγκεκριμένες ε, πολιτικές και συγκεκριμένα μέσα. Οι πολιτικές με την κατάσταση ή επανιστοχής θα, θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες τακτικές στις οποίες οπωσδήποτε πρέπει να μην ξεπερνιέται ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Ε, βεβαίως ε, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μορντού που είναι πάντα στη διάθεσή μας ε, και ανταλλάσσει πληροφορίες μαζί μας αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένας αμόντους οπεράντη ο οποίος ε, στην ουσία δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά τον δικό μας ρόλο. Εμείς χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη άρα και περισσότερη ελληνική. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών που αιτούνται διεθνού προστασία δεν είναι δυνατόν να αντιτίθενται στη να αντιτίθενται στις άτυπες ε, ε, συμφωνίες. Ε, θα πρέπει σε κάθε συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι εύκολα αναγνώσιμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαπραγματεύσεις με την Αλγερία και το Μαρόκο δεν έχουν προοδεύσει, βρίσκονται σε νεκρή φάση. Όσον αφορά την Ιορδανία, όσον αφορά άλλες χώρες της Αφρικής, επίσης, πώς εξηγείται αυτή την κατάσταση για το Αφγανιστάν Αφγανιστάν ε, θεωρεί ότι είναι ικανοποιημένη η Κομισιόν. Άλλη μια ερώτηση. Ποιε είναι οι πραγματικέ ε, εγγύσει ε, ότι οι επανεισδοχέ γίνονται σωστά και και σε σεβασμό του διεθνού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Έχουμε ανθρώπου στην Ευρώπη οι οποίοι έχουν επαναπατριστεί χωρί την διάθεση χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους ε, και ε, τέλος ε, ξέρουμε όταν αν τα άτομα αυτά φτάνοντας στις χώρες τους εντάσσονται σε προγράμματα συγκεκριμένα για να ξεπεράσουν τα ενδεχόμενα προβλήματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φανβέλτ. Ναι, βεβαίω, πολύ λογικά είναι όλα αυτά. Ε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει κάποια αίτηση και η οποία δεν έχει γίνει δεκτή να επιστρέφουν στην χώρα προέλευση τους, καταγωγή τους πολύ όμως νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι λίγο πιο περίπλοκη από αυτή που μας παρουσιάσατε. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω, όπως και η Σνάνσφος Κέγγε, είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ε, κάνουμε σωστές ε, ε, συμφωνίες επανεισδοχής με τις χώρες αυτές. Πιστεύω λοιπόν και το λέω ότι εμείς ως, έχοντας, ως έχοντες την οικονομική δύναμη μπορούμε να ασκήσουμε και πίεση. Έχουμε μοχλούς πίεση εσείς μας δώσατε μια εικόνα που όλοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και γυρίζουν πίσω αλλά στην πρακτική, στην πραγματική ζωή πώς είναι αυτό μια οικογένεια η οποία επιστρέφει στο Αφγανιστάν με παιδιά τα οποία ε, έχουν ε, περάσει πολλά χρόνια σε μια οποιαδήποτε χώρα στην Ολλανδία ή κάπου αλλού ε, κορίτσια τα οποία έχουν μεγαλώσει εδώ στην Ευρώπη και που ξαναγυρνάνε ε, στο Αφγανιστάν. Ποια ζωή τους ε, περιμένει εκεί. Η Κομισιόν ελέγχει πώς ζουν τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί. Θα συμφωνήσω με την Σιλβία. Έχουμε νομικά εργαλεία και εδώ αναφέρομαι σε μια γενική τάση. Ε, η Κομισιόν ε, ε, προσπαθεί να βρει κάποια μέτρα έτσι ώστε να, γιατί βλέπουμε ότι η Κομισιόν προσπαθεί να βρει συνέχεια λύσεις εκτός του νομικού πλαισίου. Μα το νομικό πλαίσιο όμως υφίσταται γιατί το έχουμε δημιουργήσει έτσι ώστε να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις. Εδώ μιλάμε για συμφωνίες μη, νομικά, δεσμευτικές νομικά για την επανεισδοχή. Αυτό είναι πολύ τη μόδα τώρα τελευταία. Αλλά εγώ είμαι πολύ παλιωμοδίτησα και νομίζω ότι το νομικό πλαίσιο ε, ε, έχει λόγο που έχει δημιουργηθεί και εγώ το θέλω το νομικό πλαίσιο αυτό. Ποια είναι τα ειχέγγυα λοιπόν τα οποία έχουμε. Τέλο. Τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν έτσι ώστε να ε, έχει πραγματικά νομικές συμφωνίες, πραγματικά νομικά εργαλεία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, I will equally... Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τα όσα υπόθηκαν, αλλά ε, σε ό,τι αφορά ε, τα γενικότερα σχόλια που μας θέσετε να κάνουμε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πολιτική ασύλου, ε, το ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τα υψηλά μας ε, πρότυπα, πραγματικά είναι λίγο, χειροτερεύουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι λίγο απάνθρωπες οι συνθήκες σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που κάνουμε για να μην εισέρχονται, για να τους επιστρέφουμε, λαμβάνοντα υπόψη τα όσα συμβαίνουν για παράδειγμα στην Ινδία και στη Λιβύη. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο η γενική αξιολόγηση που κάνατε είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε όλοι μα. Μετά, σε ό,τι αφορά την πολιτική επιστροφών, είπατε ότι χρειαζόμαστε μια ανθρώπινη και αποτελεσματική πολιτική επιστροφών, αλλά ουσιαστικά αυτό που είναι όλο ένα και περισσότερο είναι περισσότερο απάνθρωποι ε, και ανήθικη αυτή η πολιτική επιστροφών. Ε, και εγώ αναφέρομαι στη δική μα ε, χώρα. Έχουμε, είμαστε, έχουμε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου έχουμε νέου, οι οποίοι ενδεχομένω και άνελοι, οι οποίοι επιστρέφουν σε μια χώρα στην οποία δεν έχουν ποτέ πατήσει το πόδι τους σε μια χώρα ανασφαλή και σε μια χώρα όπου είναι ε, και, όπου έχουμε ε, κινητοποίηση από την πλευρά ε, μια σειρά των της κοινωνία των πολιτών, από πολιτικούς, από κοινότητες, προκειμένου να σταματήσει μια τέτοια πολιτική μεταφορών. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο θα μπορούσε να είναι η κοινή μα προσέγγιση εάν δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος τη γιατί εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να την εξετάσουμε, δεν μπορούμε να την αξιολογήσουμε. Οπότε θα υπάρξει μια επαναξιολόγηση. Και αν μετά από γίνει μια ε, τέτοια επαναξιολόγηση θα σταματήσει κανεί ε, τι ε, επιστροφέ. Για παράδειγμα, όπω ανέφερε συνάδελφο, σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να δεχτούμε να συνεχίζονται τέτοιου είδου πολιτικέ. Ή δεν μπορεί να υπάρξει ένα κανόνα σύμφωνα με τον οποίο δεν θα επιστρέφονται άτομα σε χώρε τι οποίε δεν έχουν ποτέ βρεθεί ποτέ στο παρελθόν. Άρα λοιπόν Νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τις ευθύνε μας γιατί προβαίνουμε σε άτυπες συμφωνίες ε, ακριβώς επειδή δεν έχουμε ε, ευθύνη για αυτές και αυτό σημαίνει βέβαια ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δυνατότητες καταχρήσεων και καταχρήσεις σημαίνουν πιο απάνθρωπες οι πολιτικές. Κυρία δεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ σε ό,τι αφορά την προσφορά που μας έγινε να λάβουμε πιο λεπτομερείς ε, πληροφορίες. Νομίζω πως αυτό είναι το δικό μας αίτημα. Ε, και η απάντηση όμως που λάβαμε ήταν ε, και πάλι μια επιστολή που περιλαμβάνεται κάποια συνοπτικά δεδομένα, όπου υπάρχει μια ε, μίξη, αν θέλετε, όλων των διαφορετικών ζητημάτων, δηλαδή στοιχεία από επίσημες συμφωνίες και μετά στοιχεία από ανεπίσημες συμφωνίες. Όταν λοιπόν μας αποστέλλετε μια επιστολή όπου μας λέτε όπου δαπανούμε 14,9 εκατομμύρια ευρώ και ε, δημιουργούμε θέσεις εργασίας στην Κάμπια, ε, αυτό δεν, είναι, δεν αποτελεί στοιχείο που μα ενδιαφέρει. Αυτό αποτελεί ζήτημα που αφορά άλλη επιτροπή. Εμεί πρέπει να προβαίνουμε στον έλεγχο αυτών των συμφωνιών επιστροφών και διαπιστώνουμε ότι όλο ένα και πιο δύσκολο καθίσταται να προβαίνουμε στον έλεγχο αυτό γιατί ακριβώ υπάρχουν όλο και περισσότερες ε, ανεπίσημες, άτυπε συμφωνίε, Οπότε ελπίζουμε να υπάρξει περισσότερη συνεργασία από τη δική σα πλευρά προκειμένου να ασκήσουμε αυτό την εξουσία ελέγχου που έχουμε και σας ξαναλέω μια άτυπη συμφωνία δεν επιτρέπει τον επίσημο έλεγχο, την επίσημη παρακολούθηση του τι συμβαίνει με κάποιον ο οποίος έχει επιστρέψει σε μια χώρα. Δεν μπορεί να προβεί λοιπόν κανείς αποτελεσματικό έλεγχο στο πλαίσιο μιας άτυπης συμφωνίας και επίσης δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος σε ό,τι αφορά την πλευρά της χώρας που λαμβάνει αυτή την επανεισδοχή. Ε, δηλαδή ε, δεν νομίζω πω στο πλαίσιο μια τέτοια ε, άτυπη συμφωνία η κυβέρνηση του Αφγανιστάν ή οποιαδήποτε άλλη χώρα του Μάλι ε, υποχρεούται να λογοδοτήσει ενώπιον του Κοινοβουλίου τη. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σαφεί γίνεται. Εσεί, για παράδειγμα, όταν μα λέτε ότι ολοένα και περισσότερε χώρε δεν θέλουν να ε, ξεκινήσουν διαπραγματεύσει σε ό,τι αφορά επίσημε συμφωνίε, νομίζω πω θα ήταν χρήσιμο για μα και να θα μας βοηθούσε σε ό,τι αφορά τον έλεγχο μας να μας πείτε ποια είναι η επιχειρηματολογία που, ζητούν που χρησιμοποιούν αυτές οι χώρες. Γιατί ε, σε, πιο μετά μας λέτε ότι ε, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ακτή του στην Κάμπια και την Κάνα τέτοιου είδους ε, συμφωνίες. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν ποιος αποφάσισε ότι πράγματι αυτέ τι χώρε δεν είναι τεθειμένε να προβούν στη σύναψη συμφωνία και κατά συνέπεια καλό θα ήταν να ξεκινήσει ε, μια διαδικασία ανεπίσημη συμφωνία. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ασκήσω λοιπόν την εξουσία ελέγχου μου γιατί δεν υπάρχουν τα στοιχεία μου για να καταλάβω πώ λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση. Και σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που μα στέλνετε, ναι, είμαι ικανοποιημένη τα στοιχεία που μα στέλνετε, αλλά αυτό το παράρτημα το οποίο αποτελεί για παράδειγμα ε, ε, τις επιστροφές σε ό,τι αφορά τις κύριες τρίτες χώρες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν περιλαμβάνονται εδώ το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μαρόκο, ο Νίγηρα, ε, το Μαλί, η Νιγηρία και η Αρκτή του Ελεφαντοστού. Υπάρχουν στοιχεία μέσα στην επιστολή σα για αυτέ τι χώρε, αλλά δεν περιλαμβάνονται εδώ στον πίνακα. Σα παρακαλώ, ε, περιλάβετε και αυτά τα στοιχεία στο παράρτημα. Μην μα λέτε πω η Μαυριτανία και η Ινδονησία αποτελούν τι κύριε χώρε που μα ενδιαφέρουν. Αναφέρομαι εδώ ενδεικτικά έτσι, σε κάποιες ε, χώρες από ένα μακρύ κατάλογο. Ένα-δυο ακόμα ε, ε, ερωτήματα θα ήθελα να θέσω, Πρόεδρε, και γνωρίζω ότι έχω περβεί το χρόνο μου. Ε, σε ό,τι αφορά την Αιθιοπία, γνωρίζω από μία πηγή. Ναι, νομίζω πως έχετε υπερβεί το χρόνο σας, συνάδελφα. Νομίζω πως... Ε, Πρόεδρο. Ε, πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε πει όλοι ε, δύο λεπτά θα μιλήσουν, έχετε ήδη μιλήσει για τέσσερα λεπτά. Ναι, ευχαριστώ, Πέρε. Σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με την Αιθιοπία, γνωρίζω ότι υπάρχει μια αξίωση από την πλευρά τη Ένωση. Η Αιθιοπία να αποδεχτεί 58 άτομα προτού γίνει περαιτέρω ε, διάλογο σε ό,τι αφορά την, τις περαιτέρω συζητήσεις σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική ε, συνεργασία. Νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό και το γνωρίζω από άλλη ανεπίσημη πηγή. Πρόεδρος. Ε, νομίζω πως υπήρχε εδώ ένα μεγάλο σπρέτσι το οποίο ε, δεν εκτυπώθηκε ολόκληρο σε αυτή τη σελίδα οπότε είναι και ευθύνη από τη δική μας πλευρά το ότι ενδεχομένως να μην περιλαμβάνονται μια σειρά από χώρες σε αυτό το πίνακα. Κύριε Κλαδίνη τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που οργανώσατε αυτήν την ε, συνεδρίαση και με μεγάλη ε, χαρά άκουσα και τις ε, πληροφορίες. Στα έγγραφα τα οποία μας στείλατε λέτε ότι η Νιγηρία παραμένει ε, η κύρια χώρα προέλευσης ε, παρατύπων ε, εισόδων. Επίσης λέτε ότι η Νιγηρία είναι η χώρα ε, που, μετράει τα περισσότερα θύματα, γυναίκες κυρίως, ε, θύματα τράφικινγκ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ε, σκέφτεστε να πάρετε κάποια επιπλέον μέτρα έτσι ώστε να βρείτε ποια είναι αυτά τα δίκτυα που εμπορεύονται ανθρώπους γιατί χρειαζόμαστε και λύσεις. Θα πρέπει όχι απλά να ανακοινώνουμε ότι έχουμε διαπιστώσει κάποια πράγματα, θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα δυνατότητα να ε, βρούμε κάποια λύση ε, γιατί οι επιστρεφόμενοι ε, στην ουσία οι επιστρέφοντες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα λόγω των δικτύων αυτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λέωνα, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστούμε πολύ κύριε Μορντή για την παρουσίασή σας. Βεβαίως το ζήτημα της επανεισδοχής παραμένει ο αδύναμος κρίκος του συστήματος ασύλου και τη μετανάστευση ε, γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι ενθαρρυντικά τα πράγματα. Πάντως ε, ευχαριστούμε που μας υπενθυμίσατε για μία ακόμα φορά ότι ε, η επανεισδοχή νομίμω διαμενόντων προβλέπεται ήδη εις την Συμφωνία του Κοτονού. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι μας. Μία, ερώτηση σε συνέχεια των όσων είπε η Σοφή Ιντβελτ. Ε, ας πούμε, η Γκάνα ε, είναι από τους μεγαλύτερους ε, δωρητές αποδέκτες αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, γίνονται διάφορες ε, συμφωνίες, ρυθμίσεις ε, μαζί τους, αλλά δεν έχουμε όμως πληροφορίες, feedback. Εμείς δεχόμαστε επομένως ότι αυτή η ρύθμιση είναι φυσιολογική εγώ νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε σε τέτοιε περιπτώσει να αυξήσουμε την πίεση μέσω όλων των εργαλείων και των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μα σε τέτοιε χώρε, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη, περισσότερο feedback όσον αφορά το τι γίνεται με του ανθρώπου αυτού. Επίση, χώρε με επίσημη συμφωνία, αναφέρατε το Πακιστάν. Ε, με εκπλήσει. Large groups of Pakistani Πήγαμε στα ελληνικά νησιά ε, το καλοκαίρι ε, και ε, είδαμε ότι υπήρχαν πολλοί Πακιστανοί για τους οποίους η απόφαση περί ήταν αρνητική και οι οποίοι όμως εξακολουθούσαν να είναι στο, στα νησιά. Δεν προχωρούσαν σε επιστροφή παρότι υπάρχει επίσημη συμφωνία με τη χώρα αυτή, με το Πακιστάν. Τέλο, κάτι βεβαίως εκτό εύρου συζητήσεω, τη σημερινή συζητήσεως τουλάχιστον. Ποια είναι αυτά τα οποία είναι απαραίτητα από την ευρωπαϊκή ε, πλευρά κατά την άποψή σα έτσι ώστε τα πράγματα να προχωρήσουν πιο ε, σωστά και έτσι ώστε να υπάρξει και αναθεώρηση της οδηγίας ε, περί επιστροφών για να προχωρήσουν καλά τα πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Μόρτιου. Ε, θα δώσω το λόγο σε δύο εκπροσώπους ε, της αντιπροσωπείας, έναν από το Μαρόκο και έναν από ε, την, Ισία. Η κυρία Καντίτζα Τζιβάνι, Τζιγιάννη μάλλον από το Μαρόκο πρώτα και ο κύριος Φαγέλ Χαλιφά μετά. Κυρία Τζιγιάννη, θέλετε να πάρετε το λόγο παρακαλώ.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 Um, Παρακαλώ πολύ τη μετάφραση τώρα, αν είναι δυνατόν, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μας έδωσε την ευκαιρία να παρέμβουμε σε ένα θέμα εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Ε, είναι οικονομικό, ε, πολιτιστικό και κοινωνικό πρόβλημα ε, η μετανάστευση. Το Μαρόκο αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, διέλευσης από μεταναστευτικές ροές και από την Ευρώπη, συγγνώμη, και από την Αφρική αλλά και από την Αιγύη Ανατολή. Ε, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την... Ε, ε, αυτό είναι ο ένας μας προβληματισμός, ο άλλος είναι και η παρακολούθηση κοινωνική κυρίως των μαροκινών πολιτών που ζουν στο εξωτερικό. Ε, και εμείς θέλουμε ε, οπωσδήποτε να, τους, να βοηθήσουμε και τους μετανάστες να ενταχθούν στην χώρα μας. Όσον αφορά τώρα ε, τις μεγάλες, τα μεγάλα διακυβεύματα, το Μαρόκο έχει προχωρήσει σε νομιμοποίηση 23.000 παρατύπων μεταναστών, οι οποίοι πλέον έχουν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, κατάρτισης, εκπαίδευση, ε, ε, επαγγελματικής ένταξη κτλ. Πράγμα που δείχνει την απόλυτη πεποίθηση και δέσμευση του Βασιλείου του Μαρόκου ε, ως προς τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης το Μαρόκο προσπαθεί να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίζει το ρόλο του χωροφύλακα λοιπόν και του προστάτη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωση. 50.000 ε, προσπάθειες ε, παράνομης μετανάστευσης ε, έχει ελέγξει το Μαρόκο και έχει σταματήσει το Μαρόκο κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ισπανίας. Επίσης ε, ε, έχει ε, σταματήσει πάνω από 80 και διέλυσε πάνω από 80 δίκτυα τράφικινγκ. Επομένως η παρουσία του Μαρόκου στους τομείς αυτούς είναι παραδειγματική. Επιπροσθέτως έχει προσυπογράψει ε, δεσμεύσεις ε, για την ε, συνολική ανάπτυξη επί τη βάση win-win με, τη, με άλλες χώρες της Αφρικής. Μη λησμονούμε ότι η Αφρική ως Ήπειρος έχει πολύ σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Πιστεύουμε πάντως ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητούνται θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν σαν αποτέλεσμα την, ε, της, ε, την ενδυνάμωση των σχέσεων ε, μεταξύ των χωρών στις δύο πλευρές της Μεσογείου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Χαλίφα θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Χαλίφα. Α, ο κύριος Καλήφα δυστυχώ, δεν είναι στην αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μορδιού για να απαντήσει. Δυστυχώ, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο πλέον στη διάθεσή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Θέλουμε να ε, απαντήσει και ο κύριος Μορδιού και στο συγγνώμη του συναδέλφου που δεν είχαν την δυνατότητα ίσω να μιλήσουν όσο ε, ήθελαν και από την κυρία Κάλε. Να προσπαθήσω να απαντήσω Καταρχήν ένα θέμα αρχής και πολιτικής επιλογής. Όποτε είναι εφικτό, είναι σαφές ότι από την πλευρά της Κομισιόν προτιμούμε σαφώς μια συμφωνία επανεισδοχής η οποία θα εξεταστεί και θα τηρεί τα σχετικά άρθρα. Μια, ένα πρόβλημα είναι όμως ότι δεν βρήκαμε πάντα τα σωστά εργαλεία για να πείσουμε τους εταίρους να συμφωνήσουν σε μια τέτοια συμφωνία. Καμιά φορά είναι ότι η διασπορά επηρεάζει πολύ τα κοινοβούλια των χωρών, ε, Επίση τα εμβάσματα παίζουν μεγάλο ρόλο και δεν μπορέσαμε πάντα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσουμε μια ενιαία ε, προσφορά που θα τους ενδιαφέρει. Πολλές φορές λένε ποιες είναι οι οδοί για την νόμιμη μετανάστευση. Η DG Home εργάζεται πάνω σε αυτό. Όποτε μπορούμε, ξεκάθαρα λοιπόν αυτή είναι η προτίμησή μας. Εκεί που δεν μπορούμε να έχουμε επίσημη συμφωνία επανεισδοχής, η νομική υποχρέωση κυρίως για πολλούς Αφρικανούς εταίρους, ήδη υφίσταται επισήμως το άρθρο 13 της Συμφωνίας του Κοτονού. Για να δούμε ποιες είναι αυτές οι άτυπες ρυθμίσεις. Καταρχήν, δεν είναι δεσμευτικά νομικά κείμενα, δεν δημιουργούν υποχρεώσεις, νομικά δικαιώματα, αν θέλετε, αναφέρουν την ε, αμοιβαία πρόθεση των δύο μερών. Για ε, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ε, αναφέρουν τον χρονικό ορίζοντα της διαδικασίας πόσο θα πάρει για να απαντηθεί έτοιμα για ταυτοποίηση, αποδεκτή τεκμηρίωση, έγγραφα, επιστροφή και με πτήσεις τσάρτερ δυνατότητα αποστολών ταυτοποίησης, δυνατότητα παρακολούθησης της αίτησης. Ε, αυτά δεν ε, είναι νομικά δικαιώματα, στηρίζονται στο άρθρο 13 της Κοτονού. Πρέπει λοιπόν να στηριχθούμε στην προθυμία της χώρας εταίρου να συνεργαστεί. Αν θεωρείτε ότι δεν έχετε τις λεπτομέρειες που θέλετε, ας κάνουμε μια ειδική συνάντηση για αυτό το θέμα. Δηλαδή να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις σας. Πάμε τώρα στις πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η κυρία Χολμάιερ νομίζω ερώτησε. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τις εκούσιες επιστροφές. Όμως έχουμε και μίνι πακέτα επανένταξης ε, μαζί με το Γραφείο Μετανάστευσης που έχουν διπλό σκοπό. Πρώτον, θα μπορέσει με αξιοπρέπεια να ε, επιστρέψει ο άνθρωπος, να έχει κάποια χρήματα για να μπορέσει να επανενταχθεί εκεί από όπου ήλθε και επίσης ε, δίνουμε και στήριξη στην κοινότητα καταγωγή προέλευσης. Υπάρχει υποστήριξη για την Αιθιοπία υπάρχει ένα μέσον για βιώσιμη και αξιοπρεπή επιστροφή με 25 εκατομμύρια ευρώ. Για το Μάλι υπάρχει ένα πρόγραμμα με 15 εκατομμύρια. Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Πακιστάν. 90 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ για τις τρεις χώρες, όλα αυτά διευκολύνουν τους ανθρώπους να επιστρέψουν και να έχουν υποστήριξη για την επανένταξη στην κοινότητά τους, γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα, τα έργα γίνονται και από τον IOM, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και ε, έχουν καλό αποτέλεσμα. Ε, άλλη ερώτηση. Ποια είναι η δυσκολία σύναψης συμφωνιών επανειζοχής με την Ισία και Μαρόκο. Το βασικό εμπόδιο που είδαμε είναι ε, η ρήτρα του υπηκόου της τρίτης χώρας που επιτρέπει σε αυτές τις χώρες να δεχτούν την επιστροφή ανθρώπων που έφυγαν από το έδαφος τους και που δεν έχουν την υπηκότητα της Τινησίας και του Μαρόκου μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη επέμεναν σε αυτό το θέμα και μάλλον θα είναι το πιο δύσκολο στοιχείο σε αυτή τη ρήτρα επανεισδοχής. Θα λυθεί στο τέλος. Θα είναι το τελευταίο που θα το λύσουμε. Τώρα, επίσης, τι ακόμα μπορούμε να κάνουμε για να υπάρχουν νομικές συμφωνίες. <clears throat> Οι αρμόδιοι υπουργοί το έχουν καταλάβει αυτό και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία ε, και στο θέμα των θεωρήσεων. Ίσως πρέπει να αναθεωρηθούν κάποια ε, ε, καθεστώτα θεωρήσεων. Βεβαίως δεν θα συμφωνήσετε αν πούμε ότι δεν θα δώσω αναπτυξιακή βοήθεια αν δεν συνεργαστείτε. Αλλά ε, θα πρέπει να δούμε τις ε, δυσκολίες με το καθεστώς, να δούμε δηλαδή προτιμησιακό καθεστώς ε, για το ταξίδι, να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση τέλος πάντων που θα μπορέσει να συγκεράσει και τις εμπορικές προτιμήσεις, αν όχι την αναπτυξιακή βοήθεια αλλά κάποια πρόσθετη βοήθεια που μπορεί να επηρεαστεί. Και έτσι μπορούμε θετικά να ευαισθητοποιήσουμε τους εταίρους ώστε να πιστούν να υπογράψουν συμφωνίες επανεισδοχής. Αυτό θα ωφελήσει όλους αναμφίβολα. Για το Αφγανιστάν κάτι που ε, βλέπουμε είναι τώρα το 30% αυτών που υποβάλλουν έτσι επιστρέφουν. Ε, για να αποφασιστεί αν θα έχουν προστασία πρέπει να δουν και τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών περιοχών στο Αφγανιστάν, γιατί είναι μερικές περιοχές πιο σταθερές από άλλες. Και αυτό είναι ένας παράγον που επηρεάζει την απόφαση που θα ληφθεί. Ομολογώ ότι δεν ξέρω καμία περίπτωση μακροχρόνιας παραμονής με οικογένεια που να ε, επέστρεψε. Ρώτησα και άλλους συναδέλφους πριν έρθω εδώ και είπαν ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν γνωρίζουν. Οι μόνες περιπτώσεις που ξέρουμε επιστροφής ε, ανθρώπων που έμειναν εδώ είναι άνθρωποι που αντιμετώπιζαν ε, δικαστικές ε, προσφυγές, δηλαδή δικαστική διαδικασία για ποινικά θέματα. Άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχουν. Η κυρία Σαρτζεντίνη το ρώτησε αυτό. Η κυρία Μπιόρκ μίλησε για το παράρτημα. Ζητώ συγγνώμη, μου φαίνεται ότι είχε πρόβλημα η διαβίβαση του εγγράφου. Είναι ε, ε, πολλά λεπτομερή στατιστικά στοιχεία εκεί για όλες τις χώρες. Θα φροντίσουμε με τη γραμματεία να το λάβετε όλοι και θα αναφέρονται και στοιχεία για τις επιστροφές και τα προβλήματα για την Αιθιοπία. Είπαμε 58 ε, άνθρωποι έχουν επιστραφεί. Δεν νομίζω ότι θα συνδέαμε αυτό με την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Πάντως θέλουμε να υποστηρίξουμε εταίρους που συνεργάζονται θετικά μαζί μας. Η ο Νίγηρ είναι πολύ σημαντικό, σημαντική χώρα ε, που συνεργάζεται καλά. Στο, κοντά στο, σε περιοχές όπως το Αγκαντέζ ε, έγιναν προσπάθειες για να τους πάρουν πίσω. Για τη διακίνηση ανθρώπων αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάλι κάναμε πάρα πολύ δουλειά με κάποιες χώρες εταίρους. Για παράδειγμα στην Ιγυρία έχουμε δημιουργήσει πλατφόρμα συνεργασίας κατά της λαθρεμπορίας ανθρώπων, την Ιγυρία. Τώρα αρχίζουμε να, κάνουμε, να συστήνουμε κοινέ ομάδες έρευνας. Ε, συνεργάζονται διοκτικές αρχές, οι αρχές επιβολής του νόμου για να ε, στοχεύσουν τους και να βρουν τους ε, διακινητές και με την Europol, την Interpol, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τη Συνοριοφυλακή συνεργαζόμεθα για να υπάρχει ροή πληροφοριών αποτελεσματική που θα πιάσει μερικούς διακινητές που εκμεταλλεύονται τους ευάλωτους ανθρώπους αδυσόπιτα. Λοιπόν, πώς προσεγγίζουμε τους εταίρους με κάθε δυνατό τρόπο. Υπάρχει νομική δέσμευση βάσει διεθνούς δικαίου. Αν πολίτης τρίτης χώρας έχει πάει παράνομα σε μια άλλη χώρα και δεν έχει ε, ε δυνατότητα να ζητήσει προστασία, θα επιστρέψει με σεβασμό στην αρχή μια επαναπροώθηση βάσει το, το χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε δυνατότητα να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και να τα προωθήσουμε όλα αυτά. Ε, αν πάρουμε το Πακιστάν για παράδειγμα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρακτικά εμπόδια και οι διατάξεις ε, μια συμφωνία επανεισδοχής δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να τεθούν σε πράξη. Καμιά φορά ε, δεν εκδίδονται από έγκαιρα τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χρειάζονται για να γίνει αναγκαστική επιστροφή ή δεν έχουν την ικανότητα οι εταίροι, δεν έχουν την πολιτική βούληση. Αν θέλουμε να είμαστε πιο σοβαροί και να, αποτε... να αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε τα... τις μεταναστευτικές ροές και να δώσουμε και προστασία με νόμιμο τρόπο, εκεί θα πρέπει να ε, αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας και θα πρέπει και κάποια κράτη-μέλη να εξετάσουν το θέμα περισσότερο. Ίσως ε, θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικότερες διαδικασίες ασύλου. Δηλαδή μεταξύ διαδικασίας ασύλου και ε, διαδικασίας επιστροφής θα πρέπει να υπάρχει ε, μια σχέση. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι άνθρωποι να φεύγουν, να συνοδεύονται κλπ. Εν περιπτώσει <clears throat> αν θέλετε λεπτομέρειες για αυτές τις ρυθμίσεις, ευχαρίστω να επανέλθω. Σοφία, ξέρω, θες να μιλήσεις πάλι, αλλά δεν έχουμε χρόνο, τι να κάνουμε. Είναι πολύ επίμαχο θέμα αυτές οι συμφωνίες επανεισδοχής ε, ε, και έχουμε άτυπες συμφωνίες και πολλές φορές παραδιάσεις προνομίων. Η, Σοφία επιμένεις, στα γρήγορα. Τι, ρω... τι θέλεις να ρωτήσεις. Όχι, είναι πολύ ενοχλητικό. Δεν απαντώνται σημαντικές ερωτήσεις. Δεν το δέχομαι αυτό. Πώς θα κάνουμε έλεγχο. Ε, Μία ερώτηση που δεν απαντήσατε είναι πώς θα εγγυηθείτε και πώς θα επαληθεύσετε ότι τα ε, πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα γίνουν σεβαστά. Και ο κύριος Λένερ το είπε. Βλέπω τον κατάλογο χωρών και δεν πιστεύω ούτε στιγμή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δυνατότητα επιρρεωής ε, σε αυτές τις χώρες, να τις πείσει για να συνάψουν μια κανονική και νόμιμη συμφωνία επανεισδοχής. Πώς γίνεται αυτό. Ε, επιτρέψτε μου να είμαι πολύ σαφής. Οποιαδήποτε επιστροφή διευκολύνεται μέσω μιας τέτοιας ε, άτυπης για παράδειγμα συμφωνίας αλλά και οποιαδήποτε άλλη επιστροφή υπόκειται σε όλα τα ένδικα μέσα προσφυγής, σε όλες τις νομικές ρήτρε και σε όλες τις αρχές του non-empowerment ε, όπω προβλέπονται σε κάθε μία από τι οδηγίε μα. Δηλαδή, κάθε μία από αυτέ τι επιστροφέ μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγή με βάση την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Και τα κράτη-μέλη τα οποία λαμβάνουν τέτοιου είδου αποφάσει θεωρούνται υπόλογα, υπεύθυνα με βάση δηλαδή την ε, νομική πρακτική που υπάρχει σε αυτά τα κράτη-μέλη. Ζητώ συγγνώμη ε, που δεν έδωσα μία τέτοια απάντηση ε, σε αυτό το λίγο χρόνο. Προσπάθησα να είμαι πολύ σύντομο και ελπίζω να σα βοήθησα. Πρόεδρος. Ναι, δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστατο για την δική μας, ε, για τον δικό μας ρόλο ε, και την ελεκτική μας ε, αρμοδιότητα. Και αντιλαμβάνομαι αυτά που ρώτησαν οι συνάδελφοι σε ό,τι αφορά ακριβώ το, το δικαίωμα ελέγχου από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση και με τι συμφωνίε με όλε τι χώρε που αναφέραμε εδώ. Ε, δεν μπορούμε να παραξετάσουμε αυτό το ζήτημα, δεν έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά ε, στο πλαίσιο των ε, ε, επαφών που είχαμε και το Σεπτέμβριο και, αυτών, και τη σημερινή επαφή, κάναμε ανταλλαγή απόψεων, αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάξαμε την άποψή μας σε ό,τι αφορά το ποια θεωρούμε πως θα πρέπει να είναι εξουσία ελέγχου από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, πάντως σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε υποκατάσταση αυτής της εξουσίας και θα γίνει μια συζήτηση ε, και σε δικό μας επίπεδο και στο επίπεδο των συντονιστών. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια, ένα τέτοιο δικαίωμα και θα ήθελα να έχουν τη δυνατότητα και στο μέλλον τα κράτη-μέλη να θέσουν ερωτήματα και σε εσά και στην Επιτροπή γενικότερα. Οπότε ευχαριστώ ε, συνάδελφοι για τα πολύ εμφαντικά ερωτήματα που θέσατε και σίγουρα επαναλαμβάνω μια τέτοια ενημερώση όπως η σημερινή δεν αποτελεί υποκατάστατο σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ελέγχου που θα έπρεπε να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τέτοιες συμφωνίες. Ευχαριστούμε πάντως για αυτή την ενημέρωση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι τα κενά αλλά σας ε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την λεπτομερή παρουσίαση. Ε, ευχαριστώ. Λοιπόν, συνάδελφοι και η κυρία Γκάλ θα αναλάβει τώρα την Προεδρία για το υπόλοιπο της ε, Μεσσίας Δεδέξης. Uh, dear colleagues, uh, συνεχίσουμε. Έχουμε δύο ακόμα ε, σήμερα στην διάταξη πρωτού ε, περάσουμε στην ψηφοφορία της, ε, στις 6 ώρα, οπότε θα πρέπει να πιεστούμε λίγο. Το επόμενο λοιπόν σημείο αφορά την δημιουργία ενός ε, συστήματος ε, πληροφοριών του ποινικού μητρώου και τη θέσπιση λοιπόν αυτού του συστήματος ε, για τον εντοπισμό των κρατών με τεθέρων πληροφορίες ποινικού μητρώου για επικοστή των χωρών και απάτηδε προς τη συμπλήρωση του έκρης. Είχε γίνει μια πρόταση για, για το 2016, η ΛΥΒΕ υιοθέτησε τη δική της εντολή τον Ιούνιο του 2016 όπου είχαμε ως εισηγητή τον κύριο Κύρκο, αλλά μετά από την ε, διάλογο που έγινε το Συμβούλιο θεώρησε πως ε, ήταν απαραίτητο να ζητήσει από την Επιτροπή μια συμπληρωματική πρόταση σε ό,τι αφορά ακριβώς την δημιουργία ενός τέτοιου ειδικού συστήματος ε, για τον εντοπισμό των σχετικών κρατομελών. Ο κύριος Εντάλτον είναι ο εισηγητής από δική μας έπλευρα. Α, όχι. Είναι, παρευρίσκεται εδώ. Μπερδεύτηκα λίγο. Οπότε κύριε Ταλτον, έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, τα κατάφερα να προσέλθω στην ώρα μου εδώ, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Άρα λοιπόν εδώ προσπαθούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο τη συνεργασία μεταξύ των κρατομελών σε ό,τι αφορά ε, τι προσπάθειε καταπολέμηση τη ε, εγκληματικότητα γενικότερα, αλλά ειδικότερα τη τρομοκρατία. Άρα λοιπόν η ανταλλαγή των πληροφοριών σε ό,τι αφορά προηγούμενε καταδίκε και ποινικό μητρό είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά ε, την ενημέρωση, σε ό,τι αφορά την μετακίνηση ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση στον τομέα τη δικαστική συνεργασία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχει και μια ε, διάκριση σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα μεταξύ πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικών τρίτων χωρών. Ε, θεωρούμε τώρα πως η πρόταση, η νέα πρόταση που έχει υποβάλει η Επιτροπή δεν αποτελεί μεγάλη ε, αλλαγή. Γιατί ούτω ή άλλω υπάρχει μια οδηγία για το έκριση η οποία καλύπτει τα περισσότερα από τα εμφυλογόμενα ζητήματα. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να τεθούν και πάλι επιτόπιτο αυτά τα ζητήματα. Όμω ε, με τη νέα πρόταση η Επιτροπή συμπληρώνει την οδηγία έκρηση, δημιουργώντα ένα κεντρικό σύστημα για τα κρατη τα οποία θα μπορούν να διαπιστώνουν σε ποια κράτη-μέλη υπάρχουν ε, πληροφορίε ποινικού μητρώου για προηγούμενε δίκε επικών τριτοχώρων και απατρίδων. Καθώ λοιπόν εδώ έχει υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Θα ήθελα να εργαστούμε ταχύτατα χωρί όμω να επιβαρύνουμε την ποιότητα τη τελική έκθεση. Οπότε θα ήθελα ο κανονισμό να ε, παραμείνει στο πλαίσιο τη εντολή που έχει λάβει το Κοινοβούλιο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά ήδη την οδηγία για το έκθεση. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι τομεί αν θέλετε, κάποια σημεία κλειδιά στα οποία έχω κάνει κάποιε τροποποιήσει ό,τι αφορά το σχέδιο τη έκθεση. Καταρχήν, θεωρώ πω είναι ε, απαραίτητο να διευρύνουμε ε, τα background checks, ε, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα παιδιά, αλλά και γενικότερα αδικήματα που αφορούν σε ευάλωτε ομάδε. Και νομίζω πω όσοι εργάζονται, για παράδειγμα, σε επαγγέλματα από τον τομέα τη υγεία, τη εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτονται. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά των κρατών μελών σε ό,τι αφορά διμερή διαβίβαση πληροφοριών ποινικού μητρώου για άτομα τα οποία ε, διαμένουν στην δική του επικράτεια, να ε, μοιράζουν αυτέ τι πληροφορίε και να εισάγουν τι πληροφορίες πληροφορίε στη δική του εθνική βάση δεδομένων. Γιατί βέβαια ένα τέτοιο σύστημα θα λειτουργήσει μόνο επί τη βάση των όσων θα τροφοδοτούν σε αυτό το σύστημα τα ίδια κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα πρέπει να αξιοποιούμε τι πληροφορίε που έχουν τα κράτη-μέλη με βάση την οδηγία. Και επίση υποστηρίζουμε ε, να γίνεται μια διαναφορά σε ό,τι αφορά την ανάγκη για εκπαίδευση σε αυτό το, το, ε, τομέα, αλλά και σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του τεκμηρίου τη αθωότητα ε, σε ό,τι αφορά αυτά τα άτομα, ειδικότερα λαμβάνοντα υπόψη ότι το, η βάση δεδομένων έκρηση για του επικόσου τρίτων χωρών δεν είναι μια τυπική βάση δεδομένων σε ό,τι αφορά ε, πληροφορίες αυτού του είδους. Οπότε ε, θεωρούμε ότι ε, και προσπαθούμε να διευκρινίσουμε ότι μια θετική απόκριση σε μια αναζήτηση μέσα σε αυτή τη βάση δεδομένων δεν θα πρέπει να υπονομεύει το δεδομένο της αρχαιότητας ή δεν θα πρέπει να αποτελεί βάση για τις διακρίσεις. Επίσης θα πρέπει η δικαίωμα πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες να είναι δίκαιο και ισότιμο για όλους και θα πρέπει να, γίνουμε, να γίνει και μια ε, σωστή αντιμετώπιση του ζητήματο τη διαγραφή. Επίση, θεωρούμε πω είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό αυτή η συνεργασία να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό θεώρησα πω είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται και ε, φωτογραφίε όπου αυτέ συλλέγονται από την πλευρά των κρατών μελών και από τη στιγμή που το σύστημα αυτό θα καταστεί λειτουργικό. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόσβαση σε αυτό το σύστημα των διαφόρων οργανισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανταπόκριση στι δικέ του αρμοδιότητε, έχω προσθέσει και την Ευρωπαϊκή Συνοριοφύλακη με βάση τα όσα εθωτήσαμε σχετική οδηγία. Το ζήτημα τώρα των υπηκών έχει συζητηθεί ήδη σε ό,τι αφορά την οδηγία ήδη και εξετάζεται αυτή την περίοδο από τα κράτη-μέλη. Εγώ από την πλευρά μου έχω κάποιε αμφιβολίε σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη και των επικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ πω ε, αυτό που θέλουμε είναι ότι ε, ήδη υπάρχει μια πλήρη συνοπτική εικόνα του, του, του, του ποινικού μητρώου και του ιστορικού πληροφοριών και του ιστορικού από την πλευρά των τόσο σε ό,τι αφορά ε, του υπηκόου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με το νέο σύστημα τόσο για του υπηκόου όσο και για του υπηκόου τρίτων χωρών. Ε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα καταλόγου αδικημάτων και σχετικών περιόδων διατήρηση των πληροφοριών, είναι ζητήματα που αφορούν τα, την εθνική αρμοδιότητα, οπότε δεν τα θίγω εγώ στην έκθεση και από εκεί και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει ένα αρμονισμένο δικαστικό σύστημα ή ένα ευρωπαϊκό αρμονισμένο σύστημα επιβολή κυρώσεων, οπότε θα πρέπει να περιορίσουμε και τι δικέ μα εργασίε στα όσα έχουμε αρμοδιότητα. Αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία μα στο μέλλον και αναμένω με ενδιαφέρον τα σχόλια των ισχυωδών εισηγητών και των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Έχω τρει συναδέλφου Ο κύριο, Ντόγιον παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ε, και τον εισηγητή για την εισαγωγή του. Βεβαίω η ιδέα καταρχήν έτσι, για να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα καταγραφής ε, των ε, καταδικών και του ποινικού μητρώου ε, θα μπορούσε να είναι καλή. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία περιέχονται στην πρόταση της Κομισιόν και που δεν έχει, επί των οποίων δεν έχει ακόμα αναφερθεί ο εισηγητής στο 3G ε, βεβαίως μπορούν να θέσουν ερωτήματα το ένα, το μία χώρα στην άλλη. Υπάρχει το σύστημα αυτό ε, και ε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και ε, με τρίτες χώρες. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση των πολιτών που είναι πολίτες υπήκοοι μιας τρίτης χώρας αλλά και ταυτόχρονα υπήκοοι μιας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως εγώ οπωσδήποτε θα ε, υποβάλω μια τροπολογία έτσι ώστε ε, να ε, βγει από το σημείο G το θέμα της διπλής υπηκότητας. Επίσης, καταδίκες καταδίκη. Ε, η καταδίκη μπορεί να είναι από, μια μικρή, από ένα μικρό πρόστιμο μέχρι ηρκτή, ε, ε, μέχρι απόφαση φυλάκισης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε κάποιο κατάλογο αδικημάτων που θα πρέπει να είναι κάπως σοβαρά, ας πούμε αυτά τα οποία μπορεί να είναι στερητικά της ελευθερίας όχι ε, όλων των ε, καταδικών οποιασδήποτε φύσης, ε, γιατί διαφορετικά θα, το βάρος του συστήματος θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επίσης, απεικόνιση του προσώπου Θυμάμαι ε, όταν συζητούσαμε ας πούμε το θέμα ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ήταν προβληματικά αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ήταν μοναδικά και μπορούσαν να ε, καθορίσουν το άτομο. Τώρα μιλάμε και για απεικόνιση προσώπου. Επίσης στο άρθρο 7 στην πρώτη παράγραφο ε, αναφέρεται ότι ε, μπορεί η διαδικασία να ξεκινήσει βάσει ε, ποινικών, ποινικών διαδικασιών και αυτό το καταλαβαίνω αλλά και άλλων διαδικασιών και δηλαδή μπορεί κανείς να έχει απλώς μια σχετική εθνική νομοθεσία και να ξεκινήσει το σύστημα εγώ νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το φορένει υπέρποζης για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο θα ήθελα επεξήγηση από τον εισηγητή ε, για τον λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ε, να ε, έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα οι διάφορες υπηρεσίες και γιατί το δικαίωμα αυτό μπορεί να επεκταθεί ακόμα και στους συνοριοφύλακες και, τους, και στην ακτοφυλακή. Επίσης ε, ε, φαίνεται να δέχεται ο εισηγητής ε, ότι όλες οι πράξεις, όλα τα στοιχεία μάλλον τα οποία προτείνει η Κομισιόν μπορεί να, είναι, να τύχουν εκτελεστικών πράξεων. Συμφωνεί με αυτό. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να είναι λογική αυτή είναι μια πρώτη γενική τοποθέτηση, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία μόλις ανέφερε και ο Ντένις Διγιάνγκ που με βρίσκουν ε, σύμφωνο. Ε, και εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα αυτά που ε, είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. Νομίζω ότι το να περάσει ένας κανονισμός ο οποίος κάνει διαφορά ανάμεσα σε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συγγνώμη, τρίτους ε, ε, πολίτες τρίτων χωρών που τυχαίνει να έχουν και ένα διαβατήριο ε, χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει αυτό να το επεξηγήσουμε και να παίρνουμε αποφάσεις και να βάζουμε, να κάνουμε κείμενα τα οποία οπωσδήποτε δεν αντιτίθενται σε αρχές οι οποίες αναφέρονται στις συνθήκες μας. Επίσης όσον αφορά τις απεικονίσεις προσώπου μπορώ να προσθέσω το εξής Εμείς ε, περιοριστήκαμε, ε, ε, είχαμε πει να περιοριστούμε στους, στα δακτυλικά αποτυπώματα, αυτό είχαμε πει τουλάχιστον στην οδηγία και νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε, να ακολουθήσουμε διαγραμμή και στον κανονισμό, δηλαδή πιστεύουμε ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι αρκετά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν θα ήθελα κι εγώ λοιπόν να συμφωνήσω με την συμπερίληψη ε, απεικονίσεων του ε, προσώπου. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί λοιπόν στην πρόταση. Επίσης υπάρχουν και κάποια ελάσσονα σημασία στοιχεία ε, επί των οποίων δεν είμαι 100% σίγουρος. Ας πούμε δεν ξέρω εάν θα πρέπει η Frontex να έχει πρόσβαση στα θέματα αυτά. Δεν είναι υπηρεσία επιβολής νόμου αλλά μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε τα θέματα αυτά ε, και περιμένω τη συζήτηση για, την, ε, για τις συμβαστικές ε, λύσεις. Κυρία Ιντβαλτ. Η Αγγέλικα Κανίμπλερ είναι σκιώδης, αλλά δεν μπορούσε να έρθει και μου ζήτησε να κάνω μια σύντομη δήλωση για το άρθρο 3. Δεν θα μιλήσω γιατί είναι ίδια με τους προηγούμενους ομιλητέ Η Κομισιόν εξήγησε στο επεξηγηματικό μνημόνιο ότι ο σκοπό είναι λυθούν θέματα ασφάλειας και να υπάρχει πιο αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων ε, ε, σε σχέση με τρομοκρατικά πλήγματα. Δεν ε, υπάρχει όμως δικαιολόγηση σε σχέση με το έκρης TCN. Εμείς δεν έχουμε πληροφορίες ούτε αποδεικτικά στοιχεία για την αξία του αποκεντρωμένου συστήματος και ούτε για το ρόλο του έκρηστης ή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, ε, αναφέρονται κάποια στοιχεία στο επεξηγηματικό μνημόνιο, αλλά δεν ε, αναφέρονται αλλού, ε, όπως ε, πιθανές ανεπιθύμητες ε, επιπτώσεις από τις διαδικασίες ασύλου πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών ενώ δεν θα υπονομεύεται η ασφάλεια που, στην οποία αποσκοπεί η πρόταση. Να προσθέσω κι εγώ δύο ερωτήσεις. Δεν γνωρίζω την έκθεση ομολογώ, αλλά ρωτιέμαι γιατί είχαμε την ίδια ερώτηση όταν μιλούσαμε για το σύστημα ενημέρωσης Schengen. Ε, καταδικαστικές αποφάσεις ε, σε τρίτες χώρες για υπηκόους τρίτων χωρών. Πώς θα κάνουμε διάκριση μεταξύ εγκλημάτων και καταδικαστικών αποφάσεων που μπορεί να έχουν πολιτικά κίνητρα. Πώς θα κρίνουμε την καταδικαστική απόφαση ε, ενός δικαστή με βάση το δικό τους ε, σύστημα. Ε, για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Οι Ολλανδικές αρχές, και αυτό αποκαλύφθηκε από τα ΜΜΕ, δεν χρησιμοποιούν τα δακτυλικά αποτυπώματα από τα διαβατήρια όπως πρέπει. Και δεν έχουμε και εξοπλισμό σε αεροδρόμια, για παράδειγμα, για να ελέγξουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Θυμάμαι τη μεγάλη φασαρία που είχε γίνει για το θέμα αυτό, ότι θα ερχόταν η συντέλεια του κόσμου. Η Ολλανδία δεν το χρησιμοποιεί καν το σύστημα για το οποίο δόθηκε τόση μάχη. Και σίγουρα και άλλες χώρες δεν θα το χρησιμοποιούν. Και αν δεν το χρησιμοποιούν, γιατί προτείνουμε τα επόμενα βήματα, τη συνέχεια αυτού του συστήματος. Δεν πρέπει να φροντίσουμε αυτά που θεσπίσαμε πριν από δέκα χρόνια και που είναι και τόσο δαπανηρά συστήματα. Δεν πρέπει πρώτα αυτά να εφαρμόζονται πριν πάμε σε άλλα. Κυρία Πρόεδρε, Μιλώ για το ΕΛΚ. Συνολικά συμφωνώ με τις προτάσεις της Κομισιόν. Θυμίζω στους συναδέλφους ότι το ΕΛΚ ήταν η μόνη ομάδα που έδωσε μάχη για το συγκεντρωτικό σύστημα τώρα είναι πλειοψηφική η άποψη αυτή και χαίρομαι. Η Frontex πρέπει να έχει πρόσβαση στο της και έχω μία ερώτηση μόνο να κάνω στην Κομισιόν. Θέλω να μάθω τη στάση της Κομισιόν απέναντι σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ηθαγένεια χώρας ε, μέλους ή άδεια παραμονής. Γιατί πιστεύω ότι το σύστημα πρέπει να επεκταθεί σε υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται εδώ ως ή μετανάστες και έχουν διαπράξει εγκλήματα. Δεν θα επαναλάβω τα άλλα τεχνικά θέματα που ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι. Η Κομισιόν Δύο λεπτά. Τρία maximum. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ε, από την πλευρά μας, από την πλευρά της Επιτροπής, ε, χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον και την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και ειδικότερα της Επιτροπής σας ε, αυτή την πρόταση η οποία βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης στο Συμβούλιο. Θεωρούμε πω πρόκειται για μια πρόταση απαραίτητη, χρήσιμη και η οποία πληρώνει ένα κενό, πληρώνει ένα κενό το οποίο υπήρχε από την αρχή τη δημιουργία του συστήματος. Ε, θεωρούμε λοιπόν πως το κεντρικό σύστημα που δημιουργούμε με αυτή την πρόταση θα πληρώσει αυτό το κενό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχόλια που έγιναν, σε ό,τι αφορά ε, τις ε, φωτογραφίες, ε, τις κατηγορίες εγκλημάτων, για τις οποίες, για παράδειγμα, θα πρέπει να πετούνται δαχτυλικά αποτυπώματα, τα ζητήματα προστασία των δεδομένων, και, τα, ε, και τις συμπληρωματικές διατάξεις, παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, παιδιών, νομίζω πω είναι ερωτήματα που θα πρέπει να απευθύνεται στο Συμβούλιο και όχι σε εμά. Οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειε εδώ. Πάντω, επιτρέψτε μου να πω ότι εμεί θέλουμε αυτό το εργαλείο να καταστεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο θα συμπληρώνει το σημερινό σύστημα ΕΚΡΙΣ, το οποίο είναι βέβαια ένα δίκτυο αποκεντρωμένο και θέλουμε αυτό το κεντρικό σύστημα να μας ε, ε, επιτρέπει να εντοπίζουμε ταχαίως το κράτος μέλος που διαθέτει κάποιες πληροφορίες ποινικών μητρώου, ώστε να γνωρίζουμε και να απευθυνόμαστε γρήγορα στο κράτο μέλο το, ε, εκείνο το οποίο διαθέτει κάποιε πληροφορίε για πει επίκο τρίτη χώρα σε άπατρη. Άρα λοιπόν αυτό θέλουμε να κάνουμε, να εντοπίσετε γρήγορα το κράτο μέλο μέσω του κεντρικού συστήματο. Το αρχικό σύστημα έκρη επιτρέπει την χρήση των ποινικών μητρών για στόχου άλλου, των ποινικών ερευνών. Άρα λοιπόν, με τέτοιο είδου ε, άλλε δικαιολογήσει υφίσταται ε, ε, ήδη. Οπότε, αν ε, υπάρχει κάποια έλλειψη στο πλαίσιο του κεντρικού συστήματο, το αν το προβλέπει ήδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, του υπηκόου ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν διπλή κωδικότητα, δηλαδή και έχουν υπηκότητα και τρίτη χώρα, απρόκειται για ένα ζήτημα εδώ το οποίο συζητούμε αυτή την περίοδο. Ε, και πράγματι υπάρχει εδώ ένα ζήτημα ω προ δηλαδή, τη δυνητική ε, διακριτική μεταχείριση που θα μπορούσε να προκύψει. Και δεν μπορώ αυτή ε, τη στιγμή να σα πω ποια είναι η λύση στην οποία θα καταλήξει το Συμβούλιο. Πάντω, ε, ε, μοιραζόμαστε μαζί σα ε, την ανησυχία σα ότι δηλαδή δεν θα υπρέ... πρέπει να υπάρχει καμία παράβαση εδώ σε ό,τι αφορά τόσο που βλέπει η συνθήκη και δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκριση σε ό,τι αφορά ε, την ισότιμη μεταχείριση ε, των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ακούσαμε την πρόταση που έγινε σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη με τις φωτογραφίες. θεωρούμε πως κάτι τέτοιο συνάδει με την εθνική νομοθεσία και πρόκειται για κάτι το οποίο ήθελε και η Επιτροπή στην ειδική της αρχική πρόταση. Επίσης, ε, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας ε, σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη του Frontox ως ε, ενός ακόμα οργανισμού ο οποίος θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο έκρηση της ΙΑΝ. Εμείς θέλαμε το Eurojust, το το EPPO να μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να καταχωρούν δεδομένα, απλώς να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Και αυτό γιατί, γιατί υπάρχει εδώ ένας στόχος αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά το Frontex δεν νομίζουμε ότι υπάρχει ένας τέτοιος λόγος. Δεν έχουμε πιστεί ότι χρειάζεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αξιολόγησης αντικτύπου, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Αντεβέλ, ναι, είχε γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου σε ό,τι αφορά την αρχική πρόταση για την οδηγία σε ό,τι αφορά τον κανονισμό υπήρξε ένα ε, λεπτομερές επεξηγηματικό σημείωμα το οποίο εμείς ε, υποβάλαμε ε, στο Συμβούλιο και ελπίζω το οποίο να λάβατε και εσείς από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Σε εκείνο το σημείωμα επεξηγούσαμε όλα αυτά τα ερωτήματα, πέραν δηλαδή της αρχικής αξιολόγησης αντικτύπου και βέβαια, βέβαια είμαστε ε, στη διάθεσή σας για να επανέλθουμε σε αυτά τα ερωτήματα στο πλαίσιο των επόμενων τριμερών διαλόγων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ε, παρεμβάσεις τους. Το πρώτο που θα μπορούσα να πω ε, γενικά είναι ότι το σύστημα λέει ότι οποτε, οποτεδήποτε έχει θετική, υπάρχει μια θετική απάντηση, ένα τότε ε, πρέπει να ζητήσεις τις σχετικές πληροφορίες από την χώρα από την οποία ήρθε η, θετική απάντηση. Αυτό σε γενικές γραμμές. Όσον αφορά τώρα συγκεκριμένα ερωτήματα, όσον αφορά άτομα με διπλή υπηκότητα, δεν προτείνω τίποτα στην έκθεση και ο λόγος είναι γιατί ε, ήθελα να ακούσω ποια είναι η αίσθηση ε, των ε, συναδέλφων γιατί εγώ προσωπικά συμμερίζομαι αυτά που είπε και ο Ντένις αλλά και ο κύριος Αλμπράιτ. Και εγώ θέλω να συμπεριληφθούν οι ε, δεν θέλω να, να μπουν ε, τα άτομα με διπλή υπηκότητα στον κατάλογο αυτό, γιατί διαφορετικά θα δημιουργήσουμε ε, δύο κατηγορίες, ας πούμε, πολιτών. Απ' την άλλη πλευρά, εάν υπάρχει ένα άτομο το οποίο έχει καταδίκη σε μια χώρα μέλος, όπου όμως έχει καταθέσει μονάχα την υπηκότητα της τρίτης χώρας, τότε, δεν, τότε ναι, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια, ε, σε μια τέτοια λίστα ας πούμε και γι' αυτό ε, ήθελα ε, να δω λίγο πώς το σκέφτονται και οι άλλοι συνάδελφοι. Επίσης στο Συμβούλιο υπάρχει η δυνατότητα, φαίνεται, να ε, προχωράνε ε, ακόμα περισσότερο και να αναφέρονται και σε άτομα τα οποία μπορεί να έχουν ε, δύο υπηκότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να ακούσω ποιες είναι οι απόψεις των συναδέλφων, έτσι ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και όσον αφορά τώρα το είδος των καταδικών, ναι δεν έχει μπει κατόφλι γιατί ε, ε, ε, είναι γεγονός ότι ένα τέτοιο όριο θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται διευκρίνηση. Όταν μιλάμε για θετική απάντηση δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα έχεις και απάντηση από το κράτος μέλος για το περιεχόμενο αυτής της θετικής απάντησης. Όσον αφορά την αναγνώριση προσώπου, συμμερίζομαι και εγώ τους προβληματισμούς που ακούστηκαν. Γι' αυτό λέμε ότι περιορίζουμε το σύστημα στις χώρες οι οποίες έχουν ήδη σε λειτουργία ε, ένα τέτοιο σύστημα και ότι δεν είναι υποχρεωτικό πάντα να χρησιμοποιηθεί ε, το ε, σύστημα αυτό. Και το βέβαιο είναι ότι, δεν, ότι θέλουμε να υπάρχει σωστή ταυτοποίηση των ανθρώπων στο σύστημα αυτό. Όσον αφορά την ερώτηση της Σοφή, να πω ότι μιλάμε μονάχα για αδικήματα ε, τα οποία έχουν ε, ε, λάβει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός της επικρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας ενδιαφέρουν οι καταδίκες οι οποίες ενδεχομένως βαρύνουν το συγκεκριμένο άτομο σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τη Europol. Η προσέγγιση ε, που ε, έχω για την Europol σχετικά με την ικανότητα της Europol να ε, μοιράζεται πληροφορίες κτλ ε, ε, συνήθως ε, η Europol κάνει κάποιες κοινέ έρευνες και εδώ έχω και κάποια πιθανά σενάρια από την Europol για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες ας πούμε εάν η Europol λάβει κάποια, κάποιες πληροφορίες για ποινικά δικήματα από την Αυστραλία για, για παράνομη διακίνηση συνθετικών ε, ε, ναρκωτικών ε, η δυνατότητα πρόσβασης σε κατάλογο σε μητρό προηγουμένων αδικημάτων θα μπορούσε να βοηθήσει ή αν έχουμε έναν Καναδό ο οποίος έχει λάβει ήδη προέγκριση ταξιδίου έστω και εάν ε, το αδίκημα το οποίο ενδεχομένως έχει διαπράξει οι ΗΠΑ δεν ε, ε, είναι σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί παρόλα αυτά η γνώση προϋπάρχοντος αδικήματος να βοηθήσει την Europol δηλαδή να δοθεί μεγαλύτερη να λαμβάνονται αποφάσεις επί τη βάση πιο σωστών πληροφοριών ε, και να πούμε ότι και η Europol και η Eurojust αποτελούν σημείο αναφοράς ε, για ε, προερχόμενους από τρίτες χώρες. Όσον αφορά τώρα την ακτοφυλακή και την συνοριοφυλακή, το ίδιο ισχύει και για αυτούς. Ε, ξέρουμε ότι οι εκπρόσωποι των και των, ε, της ακτοφυλακής ε, είναι παρόντες στα hot spots και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μητρό παλαιών καταδικών όσον αφορά τις πράξεις αν θα είναι κατεξουσιοδότηση ή ε, εκτελεστικές. Εμείς ε, δεν αγγίξαμε την πρόταση της ε, Κομισιόν όσον αφορά το θέμα αυτό. Ήθελα να ακούσω προηγουμένως τις απόψεις των συναδέλφων. Καταλαβαίνω ότι ο συνάδελφο ο Ντένις Δεγιάνγκ θεωρεί ότι θα πρέπει να μην είναι εκτελεστικές αλλά κατεξουσιοδότηση εξουσιοδότηση οι πράξεις. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό ξανά με τους συναδέλφους τους οποίους ευχαριστώ για τα όσα είπαν. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σωστά και να έχουμε μια ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά το θέμα αυτό και ευελπιστώ ότι θα έχουμε καλή συνεργασία με όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 27 Νοεμβρίου 6 το απόγευμα. Και πρέπει να πάμε αμέσως στο επόμενο θέμα. Έχουμε μόνο 12 λεπτά για το θέμα αυτό. Δίνω αμέσως το λόγο στην κυρία Γκραπίνη, η οποία είναι η συντάκτρια γνωμοδότησης για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Συνεργατικά και Ευφυή Συστήματα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που είμαι συγγήτρια, γιατί είμαι μέλος της Επιτροπής ΤΡΑΝ, που είναι υπεύθυνη. Ε, τονίζω κάποια θέματα Ε, το βλέπω μέσα από το πρίσμα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και επιμένω σε ορισμένα θέματα που αφορούν την προστασία των χρηστών. Αυτά τα συστήματα συλλέγουν και ανταλλάσσουν πολλά δεδομένα κοινά και ε, μη κοινά, ιδιωτικά. Είναι λοιπόν ε, λεπτό το θέμα. Η εφαρμογή των συστημάτων θα στηρίζεται στον γεωεντοπισμό, δορυφορικό εντοπισμό, ανεπαφικές τεχνολογίες, ε, η κολλήτολ, ηλεκτρονικά δηλαδή όλα αυτά. Κάποιες πληροφορίες που θα περνούν στα συστήματα μεταφορών είναι οι πληροφορίες που αφορούν την κυκλοφορία, τα ατυχήματα και δεν αφορούν ένα πρόσωπο συγκεκριμένα. Άλλες πληροφορίες πάλι έχουν να κάνουν με πρόσωπα που μπορεί να ταυτοποιηθούν. Είναι προσωπικά δεδομένα λοιπόν σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων. Και δεν είναι σαφές όταν ε, χειριζόμεθα τέτοια θέματα, πότε αρχίζουμε να θεωρούμε ότι πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. Τα οποία, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει σαφής, ρητή συγκατάθεση του χρήστη. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει εναρμόνιση της νομικής βάσης για την επεξεργασία των δεδομένων, διότι αυτά θα ισχύσουν για ολόκληρη την εσωτερική αγορά και οι χρήστες δεν πρέπει να θυγούν από την επεξεργασία των δεδομένων στα κράτη-μέλη. Οι χρήστες θα πρέπει να συγκατατίθενται στη χρήση των δεδομένων τους και να συμφωνούν με το σκοπό χρήσης. Επίσης δεν μπορεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέρα από την συλλογή ούτε με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους στόχους που έχουν τεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και ε, αναφέρεται σε βασικές πτυχές της ελευθερίας κίνησης ελεύθερης ε, μετακίνησης. Γι' αυτό θα πρέπει να αμυνθούμε κατά των καταχρηστικών πρακτικών. Αν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται ή χρειάζονται μόνο σε μια πρώτη αρχική φάση επεξεργασίας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ανώνυμα ή να μην συλλέγονται καν. Αυτό πρέπει να είναι δυνατόν. Αν ε, η επεξεργασία δεδομένων είναι υποχρεωτική, αυτό πρέπει να γίνεται με διαφάνεια σύμφωνα με τις διαδικασίες επεξεργασίας που επιλέγονται. Εξέτασα ε, ε, ε, σας παρουσίασα εν συντομία την έκθεση περιμένω την αντιδράσεις στις 24 Νοεμβρίου μία το μεσημέρι είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα συλλεγέντα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλο λόγο και θα έχουν ενιαία νομική βάση. Ευχαριστώ. παρακαλώ, κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την συντάκτρια της γνωμοδότησης για το έργο της που είναι μια πολύτιμη συνεισφορά ε, στο έργο της Επιτροπής Τραν. Να τονίσω και εγώ τη σημασία της αποφυγής επικαλύψεων αλλά κατάλαβα από την γνωμοδότηση ότι ξεκάθαρα αναφερόμαστε στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την ε, προστασία της ιδιωτικής ζωής ή privacy να υπάρχουν σαφείς ορισμοί για τα προσωπικά δεδομένα μόνο αν υπάρχουν και άλλες διασφαλίσεις που θα συμπεριληφθούν για τους οδηγούς, τους ε, ιδιοκτήτες, <clears throat> τους καταναλωτές στα αυτοκίνητα. Ε, ε, ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν τα πρότυπα, αλλά όχι να ε, κάνουμε επικάλυψη ε, εργασιών. Η προστασία δεδομένων είναι πολύ σημαντικό να αναφέρεται παντού, όπως επίσης και η ανωνυμοποίηση των δεδομένων σε αυτά τα διασυνδεδεμένα και αυτόνομα συστήματα και επίσης ε, υψηλά πρότυπα ασφαλείας ε, με κρυπτογράφηση. Μπορεί και εδώ να προχωρήσουμε ε, και σε θέματα ευθύνης. Με χαρά θα συμμετάσχω για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η γνωμοδότηση που ήδη είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ε, πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να ε, ελέγξουμε στο μέλλον πώς θα είναι αυτά τα αυτόνομα οχήματα. Συμφωνώ 100% ότι τα δεδομένα δεν πρέπει να ακολουθούν κατακριστικές πρακτικές, αλλά με αυτή την ευκαιρία σας καλώ να μην ε, το παρακάνετε. Μην με τα καλά στοιχεία. Κάποια στοιχεία χρειάζονται για λόγους ε, πλοήγησης, για λόγους προσαρμογής ε, και βελτίωσης της ασφάλειας και προστασίας των οχημάτων πολλές φορές δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμα, ανώνυμοποιημένα δεδομένα. Αυτό λάβετε, υπόψη, λάβετε το υπόψη σας στη γνωμοδότηση. Η κυρία Γκραπίνη για να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που δεν άκουσα τη γνώμη των συναδέλφων φιλελευθέρων και άλλων συναδέλφων. Συμφωνώ με πολλούς συναδέλφους ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε όλες αυτές τις απόψεις να τις συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότηση και στις 24 που είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών θα έχουμε μια πλήρη έκθεση η οποία αφενός δεν θα ε, επικαλύπτει ε, το έργο άλλων κανονισμών και γιατί και θα είμαστε και βέβαιοι ότι τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Ωραία. Ευχαριστώ κυρία Γκραπίνη. Η προθεσμία είναι στις 24 Νοεμβρίου, μία το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε και τέσσερα λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη των ψηφοφοριών. Καλό απόγευμα λοιπόν ξανά αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ πολύ καθίστε ήρε, ήρεμα. Θα ψηφίσουμε πρώτα απ' όλα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας την ψηφιακή ενιαία αγορά. Πρόκειται για την γνωμοδότηση του συναδέλφου Μίκαελ Μπόνι. Έχουμε και την ε, τροπολογία 6, την 27, 31, 34, 37, 40, 42, 99, 102, η τροπολογία 38 της κυρίας Βίκστρομ του κυρίου Συναδεινού 88, 89, 91, 92, 93, 141, 43, 44, 144 δηλαδή, 14, 15, 16, 18, 19, 20, μέχρι την τροπολογία 29 και μετά τροπολογίες 86 και 87. Έχουμε πολλές τροπολογίες οι οποίες έχουν αποσυρθεί. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ψηφίσουμε... Θα σας τα λέω, θα σας λέω και τις τροπολογίες ποιες έχουν αποσυρθεί. Γι' αυτό όμως ε, θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 94 της κυρίας Έρνστα. Επομένως, πρώτη ψηφοφορία θα αφορά την τροπολογία 94. Ε, κυρία Σαργεντίνη, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. Δυστυχώς δεν έχω μαζί μου την ε, ε, κάρτα μου. Προσπαθώ, ε, να μου, προσπαθώ ζήτησα να μου τη φέρουνε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, και, ο κύριος Αγγίγε. Ναι, ναι, και μένα καθοδόν είναι η κάρτα μου, να με μετράτε και μένα. Εντάξει, θα σας μετράω έναν έναν. Αλλά να μου πείτε όταν θα έρθει η κάρτα σας. Τροπολογία 94, άρχεται η ψηφοφορία. Να ψηφίσετε όμως, ε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Έχουμε τρεις συμβαστικές, οι οποίες πρέπει να ψηφιστούν unblock. block. Ε, συμβαστική 1, 2 και 3. Ψηφίζουμε λοιπόν επί αυτών των τριών συμβαστικών που θα ψηφιστούν από κοινού. 1, 2 και 3. Ψηφίζουμε. The Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 133. Τροπολογία 133 άρχεται. Τη βρήκατε, λέει η πρόεδρος τροπολογία 133, να την ψηφίσουμε τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 4, παρακαλώ, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική 4. Πέρας. Σαφώς εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία από τη Συμβαστική 5. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία επί της συμβαστικής 6. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική 7, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη τροπολογία. 134. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 134. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 135. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Α, μαζί με την 137. Βεβαίως. Από κοινού λοιπόν τροπολογίες 135 και 137 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απερίφθη. Απορρίπτονται οι τροπολογίες και 135-137. Ψηφίζουμε τώρα τις τροπολογίες 138 και 139 από κοινού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθησαν. Τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 30 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 30 επαναλαμβάνει η Πρόεδρος. Πέρας. Απερίφθη. Amendment 32. Τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απερίφθη. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 41 άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 64. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, πέρας, εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 81, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 84, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Και τελειώσαμε με τις τροπολογίες. Ε, τελική ψηφοφορία επί του τροποποιημένου κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μπόνη.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 Θα αρχίσουμε αύριο λοιπόν 8 και 4 σε κοινή συνεδρίαση με την ΕΚΟΝ. Καλό σας βράδυ. Να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε ε, και την, ε, σήμερα το ε, βράδυ, το απόγευμα μάλλον στις 6.30 στην ίδια αίθουσα ένα σύστημα, την παρουσίαση συστήματος μετανάστευσης κλπ.